afternoon. Καλησπέρα. Everybody here. Είναι όλοι παρόντες. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας, την απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών. Είμαστε στο σημείο 11 αφορά ελάχιστες απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκών τρίτων χωρών και των απάτριδων ως άτομα προσώπων χρήζουν διεθνούς προστασίας καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενο της εν λόγω προστασίας, αναδιατύπωση. Ε, έχουμε τη συνάδελφο Τζιν Λάμπερτ που είναι η συγγήτρια. Θα μας μιλήσει λοιπόν η συγγήτρια. θα αναφερθεί στις εξελίξεις όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους που διεξήχθησαν όσον αφορά τη σχετική οδηγία που αποτελεί ένα κομμάτι της, του πακέτου για το άσυλο. Τρεις τριμερείς διάλογοι έλαβαν χώρα μέχρι τώρα. Η συγγήτρια θα μας δώσει μια γενική εικόνα των εκκρεμωτήτων και μετά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εκπρόσωπος, η κυρία Γκάν, θα μιλήσει, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Η Ιωάννα Πατρέσκου, μάλιστα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αν παρίσταται, με τα χαράς να ακούσουμε τις απόψεις τους. Πρώτα απ' όλα, η εισηγήτρια, η κυρία Λάμπερτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πώς μας θυμήσατε. Έγιναν τρεις συνεδριάσεις τεμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο για να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Κάτι το οποίο είχαμε συμφωνήσει στην Επιτροπή μας και θα συνεργαστούμε στενά εγώ και οι σκιώδεις συζητητές και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μάλιστα για την συνεργασία τους και την προθυμία τους να συζητήσουμε τα θέματα για το πού βρισκόμαστε τώρα. Θα ήθελα να πω ότι προχωρούμε πολύ γρήγορα όσον αφορά το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ ανοιχτό το Συμβούλιο, ότι είναι πρόθυμο να ακούσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου και να μας δώσει όσα επιθυμούμε. Αυτό θα ήθελα. Δυστυχώς δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Και βέβαια συνηθισμένο και κανονικό είναι σε αυτή τη φάση. Έχουμε συμφωνία πενός θέματος το θέμα της ε, ανιχνευσιμότητας των οικογενειών, κυρίως αυτό σε σχέση με τους νέους. Αυτό λαμβάνει υπόψη ε, όλη τη δέσμη των μέτρων για το άσυλο και το όλο θέμα. Ε, έχουμε πολύ καλή διατύπωση επί της οποίας συμφωνήσαμε. Άλλοι τομείς που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας όσον αφορά τις τροπολογίες που υπέβαλε η Επιτροπή, το Συμβούλιο μας πρόσφερε κάποιες αιτιολογικές σκέψεις τις οποίες ε, εξετάζουμε και εξετάζουμε μία που προχωρά κάπως και καθορίζει το καλύτερο συμφέρον, το μεγαλύτερο συμφέρον για το παιδί. Θα ήταν χρήσιμο σε, σαν αιτιολογική σκέψη, αλλά θα θέλαμε να είναι μια αναφορά στις ορισμού του άρθρου 2 και πού στο κείμενο, στο διατακτικό θα αναφέρονται το, θέμα της ταυτότητας, του φύλου κλπ ε, υπάρχει μια πρόταση για αιτιολογική σκέψη, μπορούμε να την εξετάσουμε σαν ενδεχόμενο, αλλά θα θέλαμε η αναφορά αυτή να παραμείνει στο συγκεκριμένο σχετικό άρθρο. Μετά συζητάμε σε ποια θέση του κειμένου θα προσυμπεριλάβουμε και θέματα που άπτονται των παραδόσεων, των εφήμων ε, και πώς αυτά εντάσσονται τα ζητήματα στην αντιμετώπιση που θεωρείται απάνθρωπη, ε, υποτιμητική και εξετάζουμε σχετικές αιτιολογικές ε, σκέψεις, συζητούμε και κάποια άλλα ζητήματα όσον αφορά την αντιστοιχεία δικαιωμάτων των δύο ομάδων, εκείνων που έχουν την επικουρική προστασία, εκείνων που έχουν την πλήρη ε, προστασία του πρόσφυγα όσον αφορά την άδεια παραμονής. Εκεί είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί το Συμβούλιο ενώ θέλει να μειώσει τη γραφειοκρατία, και να περιορίσει τις δαπάνες εξετάζει μόνο τη διάρκεια ενός έτους ε, άδεια παραμονής για εκείνους που έχουν την περιορισμένη προστασία. Ε, άλλα επιχειρήματα που ακούμε βασίζονται στο κόστος και εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος αλλά παρόλα αυτά δεν προχωράμε και συζητείτε το θέμα. Υπάρχει ένας τομέας όμως που πιστεύω ότι ίσως καταφέρουμε εκεί να συμφωνήσουμε όσον αφορά την ε, διατύπωση διαφόρων ζητημάτων. Ένας τομέας όπου υπάρχει και διαδικαστικό θέμα είναι όσα αφορούν άλλα τμήματα της αναδιατύπωσης των μέτρων για το άσυλο. Όπως για τον κανονισμό του Δουβλίνου, Δουβλίνο 2, και τις συνθήκες υποδοχής. Πώς εκφραζόμαστε λοιπόν όσον αφορά την επικοινωνία σε μια γλώσσα εύληπτη ή που υποτίθεται ότι είναι κατανοητή και αυτό είναι κάτι που σαν ιδέα διαπνέει όλο το πακέτο. Για τα ευάλωτα άτομα να αλλάξει η διατύπωση εκεί και να πούμε αντί ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικέ ανάγκες Εκεί κάπου θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στη δέσμη των μέτρων. Τρίτον, θέμα οικογένειας, ορισμού της οικογένειας. Υπήρξαν δυσκολίες και για το Κοινοβούλιο το ίδιο. Εκεί έχουμε πετύχει συμβιβασμό, κυρίως όσον αφορά τους παντρεμένους ανήλικους, που θα έπρεπε να ποιο θα έπρεπε να είναι το καθεστώς που τους διέπει, το συγκεκριμένο καθεστώς. Αυτά είναι επιτάπη αυτά εξετάζονται από το Συμβούλιο. Ξέρουμε τη θέση μας κατά το παρελθόν, όταν μιλούσαμε για τους παντρεμένους ανήλικους που δεν συνοδεύονται από το σύζυγο ή σύζυγο και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει το Συμβούλιο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτι πρέπει να εξετάσουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο. Πώς θα προσεγγίσουμε τις διαπραγματεύσεις για να βρούμε μια λύση από αυτό. Διότι έχει συνέπειες και για άλλα τμήματα της δέσμης μέτρων για το άσυλο. Είναι θέμα διαδικαστικό που τίθεται, όπως σας είπα. Ίσως όσοι εισηγητέ θα πρέπει να δούμε τι συμφωνία μπορούμε να βρούμε σε συνεργασία οι εισηγητέ με τους Σκιώδης ίσως να καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει, διότι όποια απόφαση θα λάβουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αυτό θα έχει συνέπειες και για εισηγητέ άλλων τμήματων του πακέτου. Έχουμε την επόμενη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου την Πέμπτη. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε στα προαναφερθέντα ζητήματα. Πιστεύουμε εμείς πως και όδη συμμετείχαμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε κανονικά να συμφωνήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας με το Συμβούλιο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και κάποια θέματα που έχουν συνέπειες και αντίκτυπο και στα υπόλοιπα σημεία του πακέτου. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ. Η κυρία Πατρέσκου λοιπόν έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ για αυτή σας την έκθεση είναι πολύ ολοκληρωμένη. Χαιρόμαστε που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμα να προωθήσουν γρήγορα το θέμα. Και το ότι άρχισε να προκύπτει κάποιο συμβασμός. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι ορισμένα ζητήματα εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα, οπότε αναζητούμε μια συμβιβαστική λύση σε ό,τι αφορά ε, τον ορισμό των μελών της οικογένειας και τη σύγκληση των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Προεδρία του Συμβουλίου, θέλει να πει κάτι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Λάμπερτ για την εκθεσή της και την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ο πλευράς του Συμβουλίου και εμείς χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί. Περιμένουμε τις επόμενες συναντήσεις του τριμερού διαλόγου. Η Ουγγρική Προεδρία ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση ενδεχομένω κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Όπως είπε η κυρία Λάμπερτ υπάρχει διαφωνία σε ορισμένα ζητήματα, όμως ε, η ατμόσφαιρα είναι θετική και προσπαθούμε να βρούμε συμφωνία. Πράγματι το θέμα του ορισμού των μορφών της οικογένειας θα είναι θέμα κλειδί. Όμως και τα υπόλοιπα θέματα που έθιξε η κυρία Λάμπερτ για το συμφέρον του παιδιού και για το ε, φίλο ε, δεν είμαστε πολύ μακριά ε, από συμφωνία. Περιμένουμε με ανυπομονησία να καταλήξουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Thank you. Now, open floor. Ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής. Κυρία Χολμάιερ και μετά κυρία Ρομέρο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο κυρία Λάμπερτ. Δεν ήταν εύκολε οι πραγματεύσει που ανέλαβε και ε, προώθησε με πολύ μεγάλη επιτυχία πιστεύω και μέσα στην Επιτροπή μας την ίδια είχαμε πολλές διαφορετικές απόψεις ώρες-ώρες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε μία πρώτη οδηγία η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην ε, πρόοδο της, ε, ε, του πακέτου του σχετικού με, τις, με το άσυλο. Το θέμα λοιπόν των θεμάτων των σχετικών με τις οικογένειες ε, είναι πολύ λεπτό, είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζουμε. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσουμε χάρη και στη συμφωνία που έχουμε μεταξύ των ομάδων να ορίσουμε σαφείς όρους για την προστασία των παιδιών κυρίως, με κοινούς ορισμούς, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την ε, επαγρύπνη σε επίπεδο κρατών παιδιών, ε, τον, σε επίπεδο κρατών μελών, διότι βέβαια δεν επιτρέπεται τα παιδιά, ε, ακόμη και αν είναι ανηθαγενείς, να μην συνοδεύονται από τους γονείς τους, να μην έχουν τη σωστή μεταχείριση, να μην προβάλλονται δηλαδή και να μην προστατεύονται τα βασικά δικαιώματα των παιδιών. Νομίζω ότι και τα οι Ηνωμένα Έθνη έχουν σαφείς ορισμούς και διατάξεις για τα θέματα αυτά, τα οποία θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στο κείμενο αυτό. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για μια καλύτερη πρόοδο, γιατί εκεί αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν αρκετοί τομείς που πιστεύω χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία, αλλά πιστεύω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, ε, έστω να πείσουμε το Συμβούλιο σε κάποιε γραμμέ ε, οι οποίε θα είναι μεταξύ των θέσεων εκείνων και ημών και εύχομαι κάθε επιτυχία στη Τζιν Λάμπερτ στην προσπάθεια αυτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν πιο καλή και επακριβή ενημέρωση θέματα αυτά. Ευχαριστώ, Ρομέρο. Αυτή η οδηγία, όπως υπόθηκε, ε, συνοδεύεται από την ε, οδηγία των διαδικασιών. Οι δύο οδηγίες που προσπαθούν να ξεμπλοκάρουν το πακέτο ασύλου. Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι ε, ήταν καταστροφική σημασία στο μπλοκάρισμα του πακέτου ασύλου. Καταστροφική σημασία για την υποδοχή χιλιάδων ανθρώπων που ήρθαν από χώρες ε, όπου διεξάγονται πόλεμοι στη γειτονιά μας. Ε, την Μάλτα, την Ελλάδα, την ε, Τουρκία ή σε οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης και κέντρα υποδοχής που λειτουργούν σε, σε συνθήκες που απαιτούν την κοινή μας δράση. Ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αξίες μας, να τις υλοποιήσουμε αν δεν δώσουμε απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Και θα πρέπει να ξαναδούμε επίσης και τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ε, αυτή η οδηγία είναι μία από τις πιο σημαντικές ή από τις πρώτες του πακέτου ασύλου και αν καταφέρουμε να την ξεμπλοκάρουμε ε, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα Συνεπώς το έργο της κυρίας Λάμπερτ είναι πραγματικά πολύ αξιέπαινη. Ελπίζουμε ότι θα στεφθεί από επιτυχία το συντομότερο δυνατό για να πραγματικά αντιμετωπίσουμε αυτή την ντροπιαστική κατάσταση. Είναι προφανέ ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πως θα ικανοποιηθούν όλα μας τα αιτήματα, αλλά ακόμα και αν καταφέρναμε να συνεισφέρουμε κάτι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα ήταν πραγματικά κέρδο, έτσι ώστε το Συμβούλιο να καταλάβει ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι όνειδο για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Κυρία επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά των φιλελευθέρων θα ήθελα και εγώ και προσωπικώ βεβαίω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ την εισηγήτρια και για τι προσπάθειέ τη. Ήταν μακρά η περίοδο, δύσκολο το έργο. Συμβάλαμε όμω όλοι και ευχαριστώ και εγώ θερμά από πλευρά μου για τη συνεργασία. Είχαμε πιστεύω την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε κάποια σημεία. Επίσης θεωρώ ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνουμε και να προσπαθήσουμε τα σημεία αυτά να τα προαγάγουμε σε κόκκινες γραμμές να είναι τα σημεία αυτά στα οποία θέλουμε να βάλουμε την υπογραφή μας, με τα οποία θέλουμε να χαρακτηρίσουμε την οδηγία. Τα δικαιώματα των παιδιών πάνω απ' όλα, όπως υπόθηκε, ε, θα θέλαμε και μάλιστα να ενταχθούν όχι στις αιτιολογικές προτάσεις, αλλά στο διατακτικό του κειμένου. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αιτιολογικές προτάσεις ή σκέψεις, λοιπόν. Για να μην, υπάρχουν, ε, να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τη σημασία. Επίσης, η ισότητα των φύλων, ο ορισμός της οικογένειας, που είναι ένα θεμελιωδέστατο ζήτημα και στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για όλες τις οδηγίες εν προκειμένου, να υπάρχει ένας ορισμός κοινό και ισότιμος για όλες τις οδηγίες με, την, με ίδια διατύπωση, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα του τύπου να έχουμε μία οδηγία διαφορετικό ορισμό σε σχέση με μια άλλη. Πρέπει να είναι ή πολύ παρόμοιοι ή ταυτόσιμοι οι ορισμοί επιμένω για να μπορούμε να έχουμε ε, σωστά και καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να έχουμε και επικοδομητική συνεργασία και στο θέμα των ανηλίκων και παντρεμένων ε, νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Εύχομαι στην ε, εισηγήτρια καλή επιτυχία για την Πέμπτη, στον τριμερή διάλογο. Θα είμαι για λίγη ώρα παρούσα και εγώ και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα ώστε να το ολοκληρώσουμε ακόμη και κατά τη διάρκεια τη Ουγγρική ε, Προεδρία, πράγμα το οποίο θα αποτελούσε ένα πολύ θετικό μήνυμα, πιστεύω. Ευχαριστώ, κύριε Γκιούμ. Λοιπόν, πάνω σε αυτά που υπόθηκαν, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Τζιν για τη δουλειά που έκανε και που επιδίωξε τι συμφωνίε κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες σε ένα πακέτο για το άσυλο που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και εργάστηκε και με τις οδηγίες ε, που φορούσε αυτά τα χαρακτηριστικά για, να, για την αναγνώριση. Έχουμε όλη υποχρέωση να κινηθούμε, να βοηθήσουμε την Τζιν, να εμβαθύνουμε όσον αφορά την ορολογία και τις διάφορες έννοιες, όπως αυτό αναφέρθηκε στη διάκριση του ευάλωτου ατόμου και του ατόμου με ειδικέ ανάγκες, το διαχωρισμό. Δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο τέλος να έχουμε κείμενο που δεν θα είναι αρμονισμένα τα κείμενα μεταξύ τους, ε, διαφορετικής γενιάς κείμενα εντός του πακέτου ασύλου. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Διότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι επικίνδυνο. Και πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερος στην συνέχεια των εργασιών μας αυτό. Ο κύριος Ταβάρες, ο τελευταίος ομιλητής. Eh, ε, δεν θα απομακρυνθώ από τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Να ευχαριστήσω την κυρία Λάμπερτ για αυτή την πολύ και καλή δουλειά. Σε συνεργασία βέβαια με τους κοιοσηγητές και, τους, και τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να εστιασώ την, την, την ομιλία μου σε δύο πράγματα. Δύο συγκεκριμένα σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, διάκριση ανάμεσα σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ευάλωτα άτομα. Εγώ θα προτιμούσα τα ευάλωτα άτομα. γιατί τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ένας όρος πολύ ευρύς και ασαφής. Άλλωστε η έκθεση ευάλωτα άτομα ε, συμπίπτει με την ορολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει και σε άλλες εκθέσεις μας για τους πρόσφυγες κλπ. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό της οικογένειας και την περίπτωση των ε, παντρεμένων ανηλίκων. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά όταν επισκεπτόμαστε ε, στρατόπεδα, ε, κέντρα υποδοχής. Ε, μας λένε οικογένειες, για παράδειγμα σε ένα στρατόπεδο Παλαιστινίων στη Συρία, το οποίο είχε προβλεφθεί να κλείσει μάλιστα, μας έλεγαν ε, οι οικογένειες ότι έχουν παιδιά παντρεμένα στα 13-14 χρόνια τους. Και, θεω, και μας έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να τα αποκλείσουμε από τις διαδικασίες επανεγκατάστασης τους στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με πολύ προσοχή. Παρόλο ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν ε, αμφιβολίες και αντιρρήσεις. Ε, εμείς εδώ στην Ευρώπη δεν παντρευόμαστε 13-14 βέβαια, αλλά εκεί είναι ένα φαινόμενο αρκετά συχνό και υπάρχει κίνδυνος να χωρίσουμε οικογένειες, αν τους αποκλείσουμε. Πρέπει να δείξουμε, να δείξουμε έτσι επινοητικότητα για τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κρίζα ζώνη, τα οποία ακριβώς δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οικογένειες, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα ειδικό καθεστώς για αυτά τα άτομα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Bruns. Ευχαριστώ, κύριος Μπρόντς. Yes, we can't... δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το θέμα αυτό ότι μπορεί να εξεταστεί πέρα από το πλαίσιο το παρόν όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Πολλοί από αυτούς προέρχονται από την Τινησία. Η επανάσταση εκεί από ό,τι φαίνεται πέτυχε. Ε, το αυταρχικό καθεστώς κατέπεσε και η Τινησία έγινε πιο ασφαλής και πιο δημοκρατική. Τουλάχιστον αυτή η πιθανότητα δημιουργήθηκε. Αυτοί που ξεφεύγουν, φεύγουν από αυτή τη χώρα Φεύγουν το σκάνα από την ελευθερία και τη δημοκρατία, αυτοί που δημιούργησαν για τους εαυτούς τους. Η αλήθεια ποια είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι τούντες άσυλο, αλλά οικονομικοί μετανάστες. Το ευάλωτο των παιδιών τους που βρίσκονται σε άγνωστο περιβάλλον είναι κάτι ανησυχητικό. Αλλά η απάντηση σε αυτό είναι να αποθαρρύνουμε τον κόσμο ούτω ώστε να μην φέρνει τα παιδιά τους μαζί τους σε επικίνδυνα ταξίδια. Στην περίπτωση πραγματικών τον άσυλο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε γειτονικέ χώρε να δέχονται πολλού από αυτού. Όπου οι ετούντε άσυλο θα βρεθούν σε πιο κατάλληλο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι ξέρω κύριε Μπρόντς, οι γειτονικέ χώρες έχουν υποδεχτεί εκατοντάδες χιλιάδες ε, πρόσφυγες. Οπότε η χούφτα των ανθρώπων που έρχονται στη Γαλλία για να εργαστούν, αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Η κυρία Χολμάιερ ζήτησε να ξαναπάρει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Πολύ σύντομα θα θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον ορισμό της οικογένειας και τους παντρεμένους ανηλίκους. Μου φαίνεται από τη μια ακραίο το να υποχρεούμε να δεχθώ μια 13χρονη ως παντρεμένη και νομίζω ότι αυτό ε, έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τις παραδόσεις μας και τη νομοθεσία μας, ε, δεδομένου ότι είναι παιδιά ακόμη. Δεύτερον, θα έπρεπε ίσως να επισημάνουμε στα ότι εάν πρόκειται να αναγνωρίσουμε ε, κάτι τέτοιο ως δεδομένο, δηλαδή μια κοπέλα τόσο μικρής ηλικίας παντρεμένη, θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της ακύρωσης του γάμου. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως τα κράτη-μέλη όταν λένε ότι εφόσον υπάρχει η αναγνώριση θα έχουν δικαίωμα να έρθουν και τα λοιπά μέλη της οικογένειας και ως εκ τούτου και άλλα παιδιά θα έχουν το δικαίωμα της ε, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα αλλάζει ριζικά ε, η παρουσίαση του προβλήματος, η εικόνα του προβλήματος και βέβαια ο δικός μας τρόπος σκέψης, η δική μας νοοτροπία και ο πολιτισμός, η κουλτούρα μας δεν δέχονται ως γάμο παρά μόνο τον γάμο που έχει γίνει εκούσια. Θεωρώ δε ότι γάμος που έχει συναυθεί σε ηλικία 13 ετών είναι μάλλον αμφίβολο να έχει συναυθεί ε, με ελεύθερη βούληση του ενδιαφερομένου. Ευχαριστώ, λέει ο Η συγκέντρια παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια. Ελπίζω μεταξύ μας να τορθώσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο ίσιο αποτέλεσμα. Τα διάφορα θέματα που εθήκησαν. Ακούσαμε θέμα, αυτό για το θέμα της οικογένειας, των ανηλίκων παντρεμένων. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την Επιτροπή και γιατί προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία να λαμβάνει υπόψη όσο δυνατόν περισσότερα ζητήματα από αυτά που αναφέρθηκαν, στο βαθμό του δυνατού. Τα σχόλια δείχνουν τη σημασία που έχει να έχουμε ποιοτική διαδικασία, αποτελεσματική διαδικασία ασύλου για να είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων και τι ακριβώς συμβαίνει. Οι περισσότεροι από εμά κάτι θέλουμε να δούμε να λειτουργεί. Ευχαριστώ όσους μίλησαν για τα σχόλιά τους. Θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των θεμάτων αυτών γύρω από τους ορισμούς, να βρούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το όφελος εκείνων τους οποίους αφορούν αυτά τα μέτρα. και να ταιριάξει αυτό το νομοθέτημα με άλλα ευρωπαϊκά. Βλέπουμε που είναι οι δυσκολίες, δεν παραιτηθήκαμε όμως από την προσπάθεια να βρούμε μια λύση. Δεν παραιτηθήκαμε ακόμα και είμαι σίγουρη θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση κυρίως αν υπάρξουν και επαφές των διαφόρων ενδιαφερομένων με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. αντί να, βλέπουν μόνο, να βλέπουν μόνο τα προβλήματα, να δουν και τις λύσεις και τις δυνατότητες. Οπότε σας ευχαριστώ λέει πρόεδρος, πάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού Frontex και καλό τον εισηγητή, τον κύριο Μπούσουτιλ, να μας ενημερώσει σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μετά την ψηφοφορία προσανατολισμού που έλαβε χώρα τον Μάρτιο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα λάβει η χώρα τη Δευτέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε με το συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι οι αρχικές μου ελπίδες να κλείσει αυτό το θέμα επί Ουγγρικής ε, Προεδρίας έχουν, αρχίσει, έχουν αρχίσει να ε, υποχωρούν, να μαραίνονται. Γιατί το Συμβούλιο κάνει όλο και λιγότερες παραχωρήσεις παρόλη την επικοδομητική στάση της Προεδρίας. Γνωρίζουμε όλοι βέβαια ότι η Προεδρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 27 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού της. Αυτό περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Τώρα, να σας το δικαιολογήσω, μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τέσσερα είναι τα βασικά ε, θέματα της αναθεώρησης του κανονισμού Frontex να σας τα παρουσιάσω ένα προς ένα. Πρώτον, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για πολλούς από τους συναδέλφους εδώ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Frontex θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι θα έχει και τους μηχανισμούς για να το διασφαλίσει αυτό. Δεύτερον, ε, το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου. Είναι δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, να ζητά λογαριασμό από την υπηρεσία της Frontex. Τρίτον, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η ικανότητα της υπηρεσίας να επεξεργάζεται, μάλλον η δυνατότητα, το δικαίωμα της υπηρεσίας να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που τώρα δεν είχε. Τέταρτον, ενίσχυση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας Frontex που είναι και ο τελικός στόχος του όλου Να τα δούμε ένα προς ένα αυτά τα ζητήματα. Πρώτον, θεμελιώδη δικαιώματα. Η αρχική έκθεση περιλάμβανε ένα αριθμό τροπολογιών σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πολλές από αυτές τις τροποποιήσεις τις είχαν προτείνει οι Τελικά προτείναμε την θέσπιση ενός συμβουλευτικού οργάνου για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό της Frontex, έτσι ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να τη χάνουν πλήρως σεβασμού σε όλες τις διαστηριότητες της Frontex. Χαίρομαι να, με χαρά μου μπορώ να πω ότι το Συμβούλιο ε, δέχτηκε την πρότασή μας, ε, πρότεινε ένα πολύ επικοδημητικό κείμενο και προτείνει την δημιουργία ενός συμβουλευτικού φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον διορισμό ενός υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Frontex. Κάτι πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά ε, παραμένουν εκκρεμότητες. Μία από αυτές πιο σημαντική, οι πιο σημαντικές μάλλον, μερικές από αυτές οι πιο σημαντικές είναι εξής. Η δυνατότητα ε, οι αντικειμενικοί ε, παρατηρητές να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις της Frontex. Δεύτερον, η παρακολούθηση των διαδικασιών επιστροφής και επαναπρόθεση δηλαδή και τρίτον η δυνατότητα αναστολής των επιχειρήσεων όταν παρατηρούνται παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για αυτά τα τρία βασικά ζητήματα που ε, θα ενίσχυαν τη δημιουργία του Συμβουλευτικού Φόρουμ και, ε, ε, και, το, και τα καθήκοντα του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχουμε κάνει πρόοδο. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον δηλαδή, δημοκρατικός έλεγχος. Εδώ έχουμε προχωρήσει σημαντικά, νομίζω. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απεσιόδοξοι ως προς αυτό. Ε, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται επαρκώς εγκαίρως για τις δραστηριότητες της ε, Frontex συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων για συγκεκριμένες ρυθμίσεις με τρίτες χώρες. Επίσης θέλουμε η Frontex να είναι πιο διαφανή σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν ε, αναλάβει διάφορα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ε, την παροχή προσωπικού και εξοπλισμού στην υπηρεσία. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε και στο παρελθόν. Τρίτον, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Πήρε την γενναία απόφαση να προτείνει να δοθεί το δικαίωμα στην Frontex να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υπό αυστηρούς όρους όμως, Πρόεδρε, ε, σήμερα λαμβανόμενων περιορισμών και για το στόχο και για την ανάγκη και για την αναλογικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, έκανε αυτή τη γενναία πρόταση λοιπόν ε, και το Συμβούλιο ε, ε, έκανε μια αντιπρόταση πολύ παρόμοια με αυτή του Κοινοβουλίου. Συνεπώς αποτελεί καλή βάση για συμφωνία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη συμφωνία, αλλά νομίζω θα την πετύχουμε. Τέλος, και εδώ είναι το σημείο στο οποίο έχει γίνει μικρότερη πρόοδος, για την ενίσχυση των ικανοτήτων ε, της ίδιας της ε, υπηρεσίας δίνοντάς της μεγαλύτερη ορατότητα. Πώς δίνουμε μεγαλύτερη ορατότητα σε ένα φορέα. Μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι ο τίτλος που χρησιμοποιείται για τους συνοριακούς φορούς είναι κάτι που καταλαβαίνουν όλοι. Εμείς έχουμε προτείνει Ευρω... Ε, συνοριοφύλακες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό τον τίτλο. Οποιοςδήποτε δηλαδή ε, συμμετέχει σε επιχειρήσεις της Frontex θα έπρεπε να περιγράφεται με ένα ε, τρόπο που να δείχνει ποια είναι τα καθήκοντά του. Ε, συνοριοφύλακες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό κάνουν ακριβώς όταν δουλεύουν για τη Frontex ή με τη Frontex αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς όμως η ομάδα εργασία του, του Συμβουλίου δεν θέλει να δώσει πολιτική ορατότητα στην Frontex με αυτή την έννοια. Προτείνει, προτιμά ε, λέξεις ε, όπως λαγή ε, που είναι κενές περιεχομένου. Δεν είναι δυνατόν να ονομάζουμε κάποιους ανθρώπους λαγούς ή τα, τους υπαλλήλους μιας ενός ευρωπαϊκού φορέα λαγούς. Αυτό προκαλεί γέλοτα και επί της ουσίας, περισσότερο επί της ουσίας, μια και ο τίτλος ενδεχομένως ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τύπος, ε, δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και πιο ουσιαστικά θέματα στα οποία δεν έχουν καταλήξει συμφωνία για, ε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων της Frontex. Για παράδειγμα, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της, πόσο θα, κατά πόσο θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δικές επιχειρήσεις η υπηρεσία. Δεύτερον, αν θα πρέπει ε, ο εξοπλισμός να της ανοίγει κατά αποκλειστικότητα ε, ή από κοινού με συγκεκριμένα κράτη-μέλη, συγκεκριμένο κράτος μέλος κάθε φορά. Τρίτον, κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να δείχνουν αλληλεγγύη ε, στον, στην παροχή προσωπικού και εξοπλισμού. Πολλά κράτη-μέλη διαφωνούν με το να γίνει υποχρεωτική αυτή η παροχή. Θέλουν να αντικαταστήσουν το ε, επιτακτικό σάλ με το ε, δυνητικό μέι στο κείμενο. Συνεπώς ε, απέχουμε ακόμα από συμφωνία σε αυτό το κεφάλαιο. Άλλωστε είναι και το κεφάλαιο για το οποίο λιγότερο έχουμε συζητήσει. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά σημεία και το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σε κάθε από αυτά. Ξεκίνησα αρνητικά, αλλά θέλω να τελειώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Παρόλο ότι ε, αρχίζουν και μειώνονται γρήγορα οι ελπίδες να καταλήξουμε σε συμφωνία επί της, ε, του, κατά τη διάρκεια του Ουγγρικού εξαμήνου, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχει, έχουμε μια, ε, μια κινητικότητα με την ανακοίνωση της με την δέσμευση του Κοινοβουλίου και ενδεχομένως με τις προσπάθειες της ε, Ουγγρικής ε, Προεδρίας έχουμε μια κινητικότητα την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ε, δεν απελπίζομαι λοιπόν. Το τελευταίο που πεθαίνει είναι η ελπίδα, το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντροφε αισιόδοξε, αδιόρθωτε αισιόδοξε, για την πληρέστατη επισκόπηση. Ας δούμε αν η αισιοδοξία μας θα δικαιολογηθεί ακούγοντας το τι έχει να μας πει η Προεδρία. Ο κ. Ράντι, ένα εκπρόσωπος της Προεδρίας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Πολύ καλή εικόνα που περιέγραψε, που παρουσίασε ο κ. Μπουσετήρ τον τριμερή διάλογο, για τους διαλόγους. Πολεμάμε, το πολεμάμε ακόμα. Θέλουμε να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας, δεν παρετούμεθα. Ελπίζουμε επίσης να βρούμε λύση και εμείς ελπίζουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στην ομάδα υψηλού επίπεδου αυτή την εβδομάδα. Θα υποβληθούν τα πορίσματά του στην Κορεπέρ. Θα δούμε τι θα συμβεί και ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να συνεχιστεί ο τριμερής διάλογος υπό το φως των αποτελεσμάτων της Κορεπέρ. Είχαμε 103 τροπολογίες. Ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν να δούμε ποιες τροπολογίες ανήκουν σε ποιο άρθρο της αρχικής προτάσεως και να βρούμε επίσης τη σωστή ισορροπία μεταξύ των τροπολογιών. Η ατμόσφαιρα στους τριμερείς διαλόγους μου δείχνει ότι επικρατεί άνοιγμα και ειλικρίνεια. Αργά ή γρήγορα πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Ποτέ δεν παρετούμεθα. Και αν το Κοινοβούλιο επιθυμεί συνέχιση των τριμερών διαλόγων, ίσως να καταφέρουμε κάτι μέχρι το τέλος τη Ουγγρική ε, Προεδρίας. Να πετύχουμε πολιτικά αποτελέσματα ε, και να συμφωνήσουμε επί του κειμένου. Σας ευχαριστώ. Και άλλη αισιόδοξη στην αίθουσα. Καλό Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Ένρικ Νίλσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική προσέγγιση που ακολούθησε στον τριμερή διάλογο και για την πρόοδο που πετύχαμε τώρα. Όσον αφορά την αισιοδοξία μου μεταβάλλεται καθημερινά. Θα προσπαθήσω να σας ενημερώνω αν σας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, να εργαζόμαστε σκληρά. Σε κάθε συνεδρίαση κάναμε, σημειώναμε πρόοδο, ίσω αργότερα από ό,τι θέλαμε, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και καταλήγοντα σε θετική νότα, θα πω ότι χαίρομαι που τονίζει ο συγκεκριτή του δύο στόχου, του βασικού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από αρχή, δηλαδή ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου για τα μελιώδη δικαιώματα και ενίσχυση τη επιχειρησιακή δυνατότητα του δυναμικού. Ελπίζω να βρούμε φιλόδοξες λύσεις και συμβιβασμούς επί των δύο σημείων αυτών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι το λόγο. Ποιος άλλος επιθυμεί, εκτός από τους δύο. Τρεις. Τέσσερις. Η κυρία Κιγιούμ είναι η πρώτη. Θα μειώσω τη θερμοκρασία. Θα χαμηλώσω το θερμόμετρο. Θα αλλάξω το βαρόμετρο της αισιοδοξία. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Έδειξε ότι του αρέσουν τα δύσκολα θέματα του Μπουσατήλ και έχει καρδιά. Εγώ έχω απογοητευτεί όσον αφορά το feedback από πλευρά Συμβουλίου. Πληροφορίες μας έρχονται από εκεί και απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που θέτει ο συγγητή εν ονόμα του Κοινοβουλίου. Έγιναν πολλές προτάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και ειλικρινά για την ώρα δεν βλέπω την έξοδο από το τούνελ. Όμως νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα, όπως και στο προηγούμενο που συζητήσαμε, στην έκθεση για την οδηγία για τα επιλεξιμότητα, τα προσόντα για τους ε, πρόσφυγες κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε βασικά θέματα, θεμελιώδη δικαιώματα, δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς, το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου, ε, το θέμα της διάσωσης στη θάλασσα, των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Άκουσα προηγουμένως να λέγεται ότι ότι θα μείνει στη θέση το Συμβούλιο, το ίδιο και εμείς, ε, όσον αφορά αυτά τα θέματα. Τέλος, να πω Πέρα το ότι είναι δύσκολο το θέμα και η συζήτηση όσον αφορά την αδιατύπωση του κανονισμού Frontex είναι και μια συζήτηση που πόρα απέχει από το να είναι ουδέτερη. Και με την πάω του χρόνου και στην παρούσα περίοδο που περνά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μεταναστεύσεις, τα διαδοχικά κύματα από τι αραβικές χώρες και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να θέλουν να προχωρήσουν συζητήσεις στο Συμβούλιο βάσει των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι περνάμε μια κάπως περίπλοκη κατάσταση. Και ε, θα πρέπει να προβληθεί και να προθεθεί αυτό το εργαλείο ε, της Frontex. Ευχαριστώ κύριε Στρομ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπουσούτιλ για, το, για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία επίσης ως σκιώδεις συζητητές μαζί του. Ε, και θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εμένει στη βασική μας θέση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την ενίσχυση ε, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, θεμάτων κρισίμων δηλαδή. Δεν θα ήθελα να σας αποκαλύψω αν είμαι αισιόδοξη αυτή τη χρονική στιγμή, αν και ίσως κάποιοι θα ήθελαν να το διευκρινίσουν. Οφείλω να πω ότι πότε πότε είμαι αισιόδοξη και πότε όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, για τα αποτελέσματα νομίζω μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξο τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο. Ε, πολλές ήταν οι ε, δοκιμασίες στην αλληλεγγύη μας που έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο καιρό και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει από πλευράς Ουγγαρίας να δείξουμε ακριβώς πόσο εμένουμε στις θέσεις μας. Τα κράτη-μέλη έχουν αποτύχει ως προς την επίδειξη της απαιτούμενης αλληλεγγύης και αυτό μας απογοητεύει. Και όχι μόνο εμάς τους βουλευτές, αλλά και τους πολίτες ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν το θέμα των θεμελιωδών ανθρωπινών δικαιωμάτων, όλο το πακέτο αυτό που διαπραγματευόμαστε. Που μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης βρίσκω το να ενισχυθεί το δυναμικό της ε, υπηρεσίας Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμή δεν είχε ποτέ αμφισβητηθεί. Δεν είχε τεθεί καν προ συζήτηση. Δηλαδή, μα απασχολούσαν ε, τα θέματα τη ε, επεξεργασία δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να δεσμευθούμε στην ενίσχυση τη υπηρεσία, στην ευρωπαϊκή τη διάσταση, ω ευρωπαϊκή υπηρεσία δηλαδή. Και για άλλη μια φορά παρακαλώ το Συμβούλιο να σημειώσει πω τα κράτη-μέλη έχουν πολύ ακόμη πρόοδο στο θέμα αυτό να, ε, να επιδείξουν. Επίσης, τα σημειολογικά. Στην ορολογία, στο αν θέλουμε να συζητήσουμε με όρους ε, παράνομων ή ε, έκνομων ε, μεταναστών ή λάθρο μεταναστών. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα πρέπει η εκνομων μεταναστων η λαθρομεταναστων μεταναστων ειναι πολλα τα θεματα που πρεπει να συζητησουμε και πιστευω οτι θα πρεπει η επιτροπη μας να επιληφθεί των θεμάτων αυτών και να καταλήξουμε και σε μια στρατηγική για το πώς θα μπορούσαμε για κάθε μεταγενέστερη έκθεση τα θέματα αυτά να τα ρυθμίσουμε ε, μία και καλή και να μην επαναρχόμαστε διαρκώ με τι ίδιε συζητήσει. Και ελπίζω εν τέλει να επιτύχουμε του στόχου μα. Χωρί να μπορώ να γνωρίζω εάν αυτό θα το καταφέρουμε υπό την Πολωνική ή ακόμη υπό την ε, Ουγγρική Προεδρία. Πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν τι ε, προσευχές, και τα τάματα. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι με απογοητεύει αυτό το γεγονό ότι το Συμβούλιο μα δίνει την εντύπωση όλε χώρε ότι απορρίπτουν τι ε, τροπολογίε ε, που έχουμε από κοινό καταθέσει ω Κοινοβούλιο, όχι γιατί τι ε, θεωρούν κακέ ω προ το περιεχόμενο, γιατί φαίνεται να ε, συμφωνούμε επί της ουσίας, αλλά για λόγους μερικές φορές ακόμη και διαδικαστικούς ή υφολογικούς, το Συμβούλιο φαίνεται επιλέγει να απορρίψει τις τροπολογίες μας, πράγμα το οποίο όμως είναι μια πολιτική επιλογή και τη θεωρώ απαράδεκτη. Θα πρέπει το, κοινό, το Συμβούλιο να αρχίσει να δέχεται τις τροπολογίες μας και αυτό όχι μόνο εδώ, αλλά εν γέννη στη θεματολογία που μας απασχολεί μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν θα θέλαμε να δούμε περισσότερη πρόοδο και όχι μηδενιστικά επιχειρήματα και ε, απόρριψη των θεσιών μας. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας και πολλή συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Έρνστ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, προς τον εισηγητή καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι μας έχει βοηθήσει πολύ να ε, προχωρήσουμε συνεργατικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας τοποθέτησης, παρά σε διαφορετικές απόψεις από τις οποίες ξεκινήσαμε. Φυσικά και εγώ αισθάνομαι απογοήτευση για ότι δεν προχωρεί, δεν υπάρχει κινητικότητα από πλευρά του Συμβουλίου. Αφενός μεν έχουμε πολύ μεγάλες πιέσεις να αλλάξουμε αρκετά πράγματα από την ε, επίπεδο Frontex. Έχουμε θέματα φερρυπίν αντιμετώπιση των ε, προσφύγων που μέχρι στιγμής δεν είχαν ετηθεί. Έχουμε επίσης γενικότερα τον προβληματισμό το σχετικό με την Frontex ε, και την ανάγκη ό,τι είναι να αλλάξει, να αλλάξει σχετικά γρήγορα, να μην αναβληθεί περαιτέρω δηλαδή αυτή η αλλαγή, αυτή η αναδιατύπωση και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ε, ενώ η ομάδα μας εν γέννη, η ΓΚΟΕ δηλαδή, είναι επικριτική κατά της ε, Frontex, στέκεται δίπλα στο Κοινοβούλιο, στις θέσεις που εκφράζει το Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση αυτές. Ένα άλλο σημείο ε, θα πρέπει πιστεύω να πούμε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να διαλέξουμε τι τελικά θέλουμε. Θέλουμε να μιλήσουμε για παράτυπη μετανάστευση ή για λάθρο μετανάστευση. Γιατί η παράτυπη μετανάστευση μπορεί να μου αρέσει σαν έννοια, αλλά πάντως δεν εισάγει την ιδέα της διακριτικής μεταχείρισης όπως η λάθρο μετανάστευση, η οποία πιστεύω θα έπρεπε να καταργηθεί ως έννοια. Άρα λοιπόν προτιμώ τον όρο παράτυπη μετανάστευση. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και το Σύμφωνο να λογιστεί αυτά τα πράγματα και να προχωρήσει προς την ίδια κατεύθυνση, όχι δηλαδή με ε, απόλυτες θέσεις και αμετακίνητες. Επίσης σημαντική για μένα είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκείνων ε, που δεν ρυθμίζονται από το δίκαιο μένα, αλλά πραγματικά διαπιστώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο να δείχνει τέτοια πείσμονα συμπεριφορά στην υπόθεση αυτή, όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, όταν έχουμε να κάνουμε με ε, περιπτώσεις που πρέπει πράγματι να δώσουμε απαντήσεις και κατεπηγόντως και πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο πάντοτε να ε, μένει αμετακίνητο στη θέση του ή και να προσπαθεί να αναβάλει διαρκώ ε, την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Αυτό δεν μπορώ παρά να το, επικρίνω, να το δω επικριτικά. Ευχαριστώ κύριε Φλότο. Όλοι έχουμε καταλάβει πόσο περίπλοκε είναι οι διαπραγματεύσει. Χρειάζεται επιμονή από πλευρά του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών. Ε, Ω τώρα δεν έχουμε καταλήξει βέβαια πουθενά. Δεν ξέρω τι θα πίστευε ο Ευρωπαίος πολίτης ε, αν ε, ε, δημοσιοποιούσαμε ε, τις θέσεις του Συμβουλίου. Από τη μια μεριά του Συμβουλίου λέει πιο αποτελεσματική Frontex και από την άλλη μεριά επιθυμεί να διατηρηθούν τα πράγματα τόσο θολά έτσι ώστε να μην έτσι ώστε να συγκαλύπτονται ακόμα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν το κείμενο να παραμείνει ως έχει και η Frontex ε, να εξακολουθήσει να είναι α, τόσο διαφανής όσο σήμερα. Όλοι έχουμε συμφέρον ε, να δώσουμε στην ε, Frontex τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και τις περισσότερες δυνατές εγγύσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τη Frontex. Όταν λέμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται ένα αριθμό δικαιωμάτων, ε, προδιαγραφών κλπ, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν διαθέτουμε μηχανισμούς συνεχούς και αντικειμενικής αξιολόγησης και ελέγχου. Βλέπουμε όμως το Συμβούλιο να είναι πολύ διστακτικό. Ασφαλώς και έχει σημειωθεί πρόοδος, το πακέτο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως το ονομάζουμε, ε, ε, έχει κάνει κάποιο δρόμο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ελέγχου και των μηχανισμών που θα παρακολουθούν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι αξιόπιστος και διαφανής, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η Frontex και οι δραστηριότητες της ε, θα τηρούν τις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε θέσει. Αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα. Ένα κομμάτι του παιχνιδιού παίζεται και στον δημοκρατικό έλεγχο και στο κεφάλαιο του δημοκρατικού ελέγχου. Έχουμε ψηφίσει τον προπολογισμό της υπηρεσίας αυτής, οπότε έχουμε απαιτήσει να γνωρίζουμε τι συμφωνίες υπογράφει, για τη φύση των επιχειρήσεων επίσης που σχεδιάζει, ε, για τις ε, αναλύσεις κινδύνου, τις οποίες προβαίνει κλπ. Αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Νομίζω ότι εμείς θα είμαστε επίμονοι Βλέπω ε, και τη διάθεση του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών και νομίζω ότι το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο πια να ε, κάνει ένα βήμα υπέρ προς την κατεύθυνση του ελέγχου, του δημοκρατικού ελέγχου, της διαφάνειας και των εγγύσεων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής πριν επιστρέψουμε στον εισηγητή, Uh, η Frontex αναμφίβολα θα πρέπει να μεταχειρίζεται όλους και τους υπόπτους ε, ότι είναι παρανομετανάστες με την ίδια αξιοπρέπεια. Χωρίς όμως αυτό να παρακολεί το βασικό σκοπό της ε, Frontex που είναι ε, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης όταν εντοπίζονται παρανομετανάστες στη θάλασσα ή σε πλοία, ε, σε σκάφη, θα πρέπει να διασώζονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όμως, αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι, σώζοντάς τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει και την υποχρέωση, μια υποχρέωση να τους δεχτεί που δεν είχε προηγουμένως. Αυτό θα είναι σαν να ανταμείβουμε την προσπάθειά του να μπουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, τελευταίο σχόλιο. Αν θα χρησιμοποιούμε τις λέξεις ε, παράνομο ή λαθρομετανάστες ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να διαλέγει τη, δική, τη δική του ορολογία. Γιατί οι, όροι που χρησιμοποιούμε ε, έχουν ε, συνοδεύουν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν μπορούμε κανένα να υποχρεώσουμε να αντιμετωπίζει τα πράγματα και να τα σκέφτεται με το δικό μας τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ως ιδιαίτερους συναδέλφους, τους Σκιώδης και τα άλλα μέλη που συμμετείχαν στην σημερινή συζήτηση και όλος ιδιαίτερος τους σκιώδεις με τους οποίους είχα άκρος θετικές και επικοδομητικές σχέσεις εργασίας τους τελευταίους μήνες για να καταφέρουμε να καταλήξουμε ε, σε θετική κατάληξη όσον αφορά το πολύ δύσκολο θέμα. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, πάμε για τον τέταρτο τριμερή διάλογο τη Δευτέρα και αυτή η συνεδρίαση της Δευτέρας είναι πολύ σημαντική, θα είναι το κλειδί, διότι ανάλογα με τα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα ανάλογα με το πόσο θα μετακινηθεί από τη θέση του Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό, θα γνωρίζουμε κατά πόσο αυτό το χαρτοφυλάκιο θα έχει οριμάσει πλέον για να καταλήξουμε σε τελικά αποτελέσματα επί Ουγγρικής Προεδρίας. Όπως ήδη είπατε, ελπίζουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά τελικά Αυτά είναι και στα χαρακτηριστικά της διαδικασίας συναπόφαση. Συναπόφαση συνεπάγεται ότι δύο θεσμικά όργανα και όχι ένα αποφασίζουν. Ε, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Συμβούλιο να εκτιμήσει πλήρως αυτό το χαρακτηριστικό στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα γίνει τη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε φτάνουμε στο σημείο 13 της ημερήσιας ε, διάταξης έχουμε μια παρουσίαση μιας ε, μελέτης ε, του καθηγητού Dirk Van Hoel Σας ζητώ συγγνώμη που περιμένα, περιμένατε κάνα δύο λεπτά. Θα γίνει μια παρουσίαση λοιπόν σχετικά με τη μελέτη που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Πολιτικής Γάμα για το θέμα της εφαρμογή αρχή αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων στι τομεί των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και τη ε, μετανάστευση. Έχετε λοιπόν ε, το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε που αφορά το άρθρο 80 της TFU, e όπως ε, θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό το άρθρο το άρθρο 80 τη Συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νέα διάταξη, είναι μια διάταξη που είναι πολύ ευρύτερη από το κλασικό μηχανισμό κατανομής των βαρών, που είναι κάτι πολύ γνωστό σε θέματα ασύλου και ασχολείται με περισσότερο και με άλλα θέματα, όχι μόνο το ασύλο, άλλα θέματα μεταναστευτικά και μεθοριακού ελέγχου. Στη μελέτη λοιπόν εξετάσαμε τους λόγους για τον επιμερισμό των ευθυνών και υπάρχουν τρει βασικοί λόγοι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και όταν ε, υιοθετείται, θεσπίζετε νομοθεσία και προβλέπονται δράσει. Ε, είναι ένα είδο ασφάλιση λοιπόν το κίνητρο τη στιγμή όταν, όταν κυμαίνονται οι μεταναστευτικέ ροέ και το κόστο, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που θα σταθεροποιεί το κόστο και να επιτυχάνει σταθεροποίηση και να μοιράζεται το κόστος. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μειώνοντας το συνολικό κόστος το οποίο σχετίζεται με, την, με τις μεταστευτικές ροές ή κατανέμοντας αυτό το κόστος ε, με δικαιότερο τρόπο μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, πρώτο στόχος, δεύτερος στόχος για την κατανομή των ε, ευθυνών και επιμερισμού του βάρους είναι να αποφευθεί η επιβλαβής μονομερής δράση και ε, μια κατοφ θερή πορεία όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστου. Αν το κόστο μεγάλο, ίσω ένα κάτω μέλο να επαναφέρει εσωτερικού ελέγχου των συνόρων ή να στερεί κάποιου μετανάστε από κοινωνικά δικαιώματα στην επικράτεια. Αυτό να οδηγήσει σε κάποιε συγκρούσει που ίσω να θεωρούνται κάτι ανεπιθύμητο. Μετά, τρίτη προοπτική ε, είναι μια ευρύτερη, ευρύτερη στοιχεία που αφορούν την αλληλεγγύη και την αμοιβαία συνεργασία. Ποια είναι η κεντρική ιδέα, ότι εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα κυρίω όσον αφορά τι χώρε και τι περιφέρειες που είναι πλέον ευάλωτε όσον αφορά ε, τη μετανάστευση. Λοιπόν, τώρα βλέποντα κάποιε θεσμικέ πτυχέ, ε, βλέπουμε από την έρευνα ότι οι νομικές συνέπειες του άρθρου 80 είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από τις διάφορες εφαρμογές ε, πολιτικής. Οι περισσότερες από αυτές τις ε, εφαρμογές πολιτικής αφορούν άμεσες κρίσεις, απαντήσεις άμεση κρίση. Η αλληλεγγύη ε, καθορίζεται πολύ χαλαρά και αόριστα, δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το τι αποτελεί αλληλεγγύη, περί τίνος πρόκειται και Κάποιοι είπαν ότι αν θέλετε να καθορίσετε την αλληλεγγύη και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, θα πρέπει να εξετάσετε τους διάφορους στόχους και τους διάφορους στόχους τους βλέπετε στα άρθρα, 77-79 της συνθήκης και διαφέρουν. Ένα άρθρο εξετάζει τον έλεγχο όσον αφορά τα σύνορα και άλλο αφορά την υποδοχή και την παροχή προστασία όσον αφορά το άσυλο. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατορίσει κανεί την αλληλεγγύη εντό των διαφορετικών αυτών τομέων. Υπάρχουν και διαφορέ απόψεων μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα. Το άρθρο 80 ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή επίση είναι εφαρμοστέο και στα κράτη-μέλη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών και είναι μια έννοια που θα πρέπει να προσεγγιστεί πανευρωπαϊκά, όλοι να συμμετέχουν. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει διμερείς δράσεις, μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολυμερείς δράσεις. Είναι πολύ ασαφής η πρόθεση. Το ίδιο όσον αφορά τον την υποχρεωτική εθελοντική συμμετοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές όσον αφορά την εκτίμηση του θέματος από τους διάφορους φορείς του τομέα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε κάτι που είναι σημαντικό σχέση μεταξύ αλληλεγγύης και συνεργασίας, αυτό από τη μια μεριά, εμπιστοσύνης και πίστης, αν θέλετε, από την άλλη. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ευρωπαϊκό χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα και αν θέλουμε να θεωρούμε ότι λειτουργεί ο χώρο, ελάχιστο όρο για την εμπιστοσύνη ότι τα κράτη-μέλη είναι πιστά όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε να υπάρχει εμπιστοσύνη, να υπάρχει πίστη, συμμόρφωση από τα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη για να είναι πιστά στην νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντικό από καιρού καιρών η αλληλεγγύη να παίξει ένα ρόλο. Χωρί την αλληλεγγύη, καμιά φορά σε ιδιαίτερε περιστάσει είναι αδύνατον τα κράτη-μέλη ακόμα και να είναι πιστά να συμμορφώνονται ακόμα και όταν θέλουν. Η αλληλεγγύη αντισταθμίζει την έλλειψη πίστης και συμμόρφωσης. Τόσο ό,τι αφορά τα εργαλεία, αναλύσαμε διάφορα εργαλεία, τα μελετήσαμε, νομοθεσία για παράδειγμα, η ελάχιστο τουλάχιστον θα πρέπει να είναι για παράδειγμα ότι η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη αλλά αυτή η εφαρμογή ίσω δεν επαρκεί από μόνη τη έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αλληλεγγύη και πίστη εντάξει των κρατών μελών. Ε, θα ε, συζητήσαμε και το θέμα τη γενικότερη μείωση και ε, πιο ισότιμη κατανομή των του κόστους, αλλά έχουμε πολύ λίγα αριθμητικά στοιχεία, οπότε χρειάζεται να εμβαθύνουμε θα πρέπει να δούμε και τα άμεσα και τα έμεσα κόστη ε, που συνδέονται με αυτή την πολιτική. Επίσης, ε, συμφωνούμε ότι ένα βασικό στοιχείο της αλληλεγγύης είναι τα ταμεία. Τα ταμεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όμως ε, και τα κονδύλια που περιλαμβάνουν είναι πολύ μικρά και έχουν πιο πολύ το χαρακτήρα του κινήτρου, όχι της αποζημίωσης. και μπορώ να πω ότι είναι και γραφειοκρατική η λειτουργία τους. Ε, ίσως και ε, πέραν της χρηματοδότησης θα ήταν πιο σημαντική βοήθεια σε, με πρακτικούς όρους, για παράδειγμα βοήθεια στην ενσωμάτωση κλπ. Επίσης, υπηρεσίες όπως η Frontex ή η ASO ε, είναι πολλά υποσχόμενος τρόπος για το μέλλον. Όμως ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, προσωπικό και χρηματοδότηση και αυτές. Ε, ίσως ε, θα ήταν μελετήσαμε επίσης την πιο, την, το, ένα σύστημα στο οποίο θα γινόντουσαν πιο κεντρικά, θα σχεδιόντουσαν πιο κεντρικά οι επιχειρήσεις, ε, αλλά ε, δεν μας εκπλήσει το συμπέρασμα ότι η αλληλεγγύη σημαίνει περισσότερη αποκέντρωση. Η γεωγραφία επίσης ε, θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερη αξία, να τονιστεί περισσότερο, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε και τα προβλήματα και να αναπτύξουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Εξαιτία της γεωγραφικής τους, τους θέσης, το βάρος σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ περισσότερο από, ότι σε, ε, από το βάρος άλλων κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε και πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις στην ανάλυση μας, στη μελέτη μας. Ε, ξεκινώντας από τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, αναγνωρίζουμε ότι η ανάγκη για αλληλεγγύη απορρέει από την πραγματικότητα της, του οικοδομήματος της Σέγγεν και η διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή. Ε, παρόλο που ε, τώρα μιλάμε πιο πολύ για τον έλεγχο της περιοχής γύρω από τα σύνορα. Η εσωτερική ασφάλεια μπορεί να τύχει εγγυήσεων μόνο με ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης αναγνωρίζουμε όμως ότι η αλληλεγγύη σχετίζεται, σχετίζεται επίσης και με άλλους τομεί και με άλλες περιοχές, ε, όχι μόνο με τα σύνορα. Δηλαδή σχετίζεται επίση και ε, με την ε, υποδοχή, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ετώντες άσυλο. Είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη που χρειάζεται στην υποδοχή με την αλληλεγγύη που χρειάζεται στον έλεγχο των συνόρων. Ε, γενικά το έργο της Frontex είναι αξιέπαινο, αλλά έχουμε και εδώ προτάσεις, περισσότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα, επιχειρησιακό τομέα, και σε ό,τι αφορά την κάλυψη πραγμάτων τα οποία δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, ε, χορήγηση εγγράφων σε άτομα τα οποία έρχονται χωρί ταξιδιωτικά έγγραφα. Ε, σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτουμε, ε, είναι ανεπαρκή πρώτον. Δεύτερον, χρειάζεται, ίσως χρειαστεί χρηματοδότηση για την πρόσληψη προσωπικού και ίσως θα χρειαστεί να βοηθήσουμε ιδιαίτερα ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία ε, έχουν πολύ μεγαλύτερο βάρος και συνεπώς ε, πολύ μεγαλύτερο κόστος στη δράση τους. Επίσης είναι σημαντικό να αποφύγουμε ε, μονομερείς δράσεις για παράδειγμα την επιστροφή σε εσωτερικούς ε, σε έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα ε, στην ε, περίπτωση έλλειψης αλληλεγγύης, γιατί αυτό δημιουργεί σημαντικά μη χρηματικά κόστη επίσης. Επίσης, η μεταφορά προσωπικό από ένα κράτος μέλος σε άλλο ίσως είναι χρήσιμο για το ίδιο, χρήσιμη για το ίδιο το προσωπικό και τους βοηθάει να προσαρμοστούν και να καταρτιστούν. Σε ό,τι αφορά το άσυλο και την προστασία, Χρειάζεται καλή σωστή εφαρμογή ε, της νομοθεσίας για το άσυλο που ισχύει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε αυτό το κεφάλαιο. Η αλληλεγγύη μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν ε, ένα αριθμό κρατών μελών ή όταν συνδέονται με ένα παγκόσμιο βεληνικούς ε, γεγονός ανθρωπιστικής φύσεως. Ίσως είναι προβληματικό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, ζητούν περισσότερη αλληλεγγύη από άλλα κράτη-μέλη, ιδιαιτέρως όμως όταν τα ίδια αυτά δεν τηρούν τις δικές τους υποχρεώσεις. Αν λοιπόν ένα ένα κράτος-μέλος ε, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, πώς μπορεί να ζητάει αλληλεγγύη, είναι κάτι που συμβαίνει ε, και είναι αντιφατικό. Θα πρέπει να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους πρώτα το Δουβλίνο μπορεί να απαιτήσει αποζημιώσει ή διορθώσεις, διορθώσεις εννοώντας, ε, μιλώντας διορθώσεις εννοούμε για προσωρινή αναστολή, ενώ ως αποζημιώσεις εννοούμε την επανεγκατάσταση. Η επανεγκατάσταση είναι πιο κατάλληλη για τους ε, πρόσφυγες, οπότε η αλληλεγγύη εκεί θα πέσει πιο πολύ στο, στο κεφάλαιο της ε, ε ενσωμάτωσης γιατί κάποια μέλη που έχουν πολλούς ε, πρόσφυγες ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξής τους στις τοπικές κοινωνίες, οπότε ίσως χρειάζεται να, να βοηθηθούν με ένα ε, σύστημα επανεγκατάστασης. Άλλα εργαλεία θα μπορούσαν να καλύψουν καλύτερα τους ετούντες άσυλο. Για παράδειγμα, από κοινού επεξεργασία ε, των αιτήσεων, παρόλο που υπάρχουν θέματα εθνικής κυριαρχίας σε αυτό το ζήτημα. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη-μέλη που ζητούν επανεγκατάσταση ετούν τον άσυλο, ε, δεν τηρούν τις δικές σου υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το ίδιο κεφάλαιο. Βέβαια υπάρχουν γεωγραφικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να απαιτήσουν ορισμένα κράτη-μέλη ε, να βοηθηθούν διότι δεν μπορούν να διαχειριστούν ε, τον αριθμό των αιτήσεων που φτάνουν. Ε, σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση έχουμε δύο δυνατότητες που προτείνουμε. Ε, όταν υπάρχει θέμα χωρητικότητας σε ένα κράτος ε, μέλος, αυτό το κράτος μέλος ε, ε, θα μπορούσε να αναλάβει το 30% των, 30% ε, των ετούντων παραπάνω από ό,τι είχε δεχθεί το, το προηγούμενο έτος και το υπόλοιπο 70% να επανεγκαθίσταται. Αυτό ίσως είναι μια κοινώς αποδεκτή λύση. Σε ό,τι αφορά δε την ενσωμάτωση, την ένταξη, ε, και πάλι όταν ε, ο αριθμός ε, των προσφύγων ξεπερνάει τις δυνατότητες μιας χώρας θα μπορούσαν να επανεγκαθίστανται. Το κοινοβούλιο το ίδιο βέβαια είχε ζητήσει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για αναδιανομή των προσφύγων. Αυτή τη στιγμή βραχυπρόθεσμα ίσως θα ήταν σημαντικό να σκεφτούμε το σύστημα της ε, προσωρινής προστασίας, ε, αν αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί η κρίση στη Λιβύη, αυτό βραχυπρόθεσμα. Δεύτερο, ε, να δώσουμε βοήθεια στις γειτονικές χώρες, για παράδειγμα στην Αίγυπτο και στην Τινησία στην περίπτωση της Λιβύης. Ίσως θα ήταν και αυτό μια λύση και μια έκφραση αλληλεγγύης τρίτο στοιχείο, και έτσι επιστρέφουμε στις παλιότερες πολιτικές του 80 και του 90, να εργαστούμε σε πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα επανεγκατάστασης σε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Εδώ η αλληλεγγύη δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και δεν μας εκπλήσει αυτό. Ίσως είναι σημαντικό να πηδηχθεί η αλληλεγγύη και εδώ, διότι όταν, έχουμε μια, όταν αποτυχάνει η μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας μπορεί αυτό να επηρεάσει και άλλους τομείς. Γιατί αν κάποιος ε, δεν μπορεί να γίνει δεκτός ως μετανάστης μπορεί να ζητήσει άσυλο για παράδειγμα. Η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού όμως δημιουργεί προβλήματα, είναι πολύ προβληματικό να εξασφαλίσουμε τη συμφωνία όλων των κρατών μελών για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική του εργατικού δυναμικού. Ο ανταγωνισμός δεν θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια σίγουρα, οπότε ε, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε δεν θα μειωθούν στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τι θεωρίε, δεν έχουμε πολλά προβλήματα, σε ό,τι αφορά την ένταξη δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο το, ε, δεν θα πρέπει να βλέπουμε το εθνικό επίπεδο, αλλά το τοπικό επίπεδο. Γιατί οι προσπάθειε σε πολλά κράτη-μέλη είναι σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Και εκεί οι ανάγκε αυξάνονται εξαιτία ε, περικοπής, ε, δημοσιονομικών περικοπών σε πολλά κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εργαστούμε επί μια αποζημίωση, αντιστάθμιση όταν έχουμε προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή, και την επαναπρόθεση. Ε, έχουμε ε, περισσότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης ε, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική, τη διαβίας παρά την εθελούσια επιστροφή με κοινέ πτήσεις και συμφωνίες επανεισδοχής. Τώρα, πού θα μπορούσαμε να δείξουμε αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τους νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς. Ε, έχουμε αφιβολήσει ό,τι αφορά την συλλογική σταθερότητα ε, και των σχέσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων. Εκεί θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Θα μπορούσαμε επίσης να σε επίπεδο ε, νομοθεσίας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την παράνομη μετανάστευση. Με την, επίσης με την πολιτική, την αναπτυξιακή μας πολιτική θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε το εμπόριο, το εμπόριο ανθρώπων με την ενσωμάτωση. Και στην ενσωμάτωση επίσης είναι δύσκολο να δούμε πού θα μπορούσαμε να ε, δείξουμε αλληλεγγύη. Είναι δύσκολο ο υπολογισμό του κόστους. Ε, ε, είναι δύσκολο αποζημιώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, την, ε, ή τα κράτη-μέλη να έχουν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τοπική ένταξη. Να φτάσω στα συμπεράσματα. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό για κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκεφτόμαστε το κατά να απαιτείται ελεγγύη. Αυτό το αναφέρει το άρθρο 80 αλλά είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς, σε κάθε βήμα που θα κάνουμε. Αν απαιτείται αλληλεγγύη, τότε τα ε, εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να, εξασφαλ... να αποφασίζουν αν ε, η αλληλεγγύη αυτή θα είναι θελοντική και αν ναι, ποιοι θα συμμετάσχουν, αν θα είναι ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αν θα είναι απλώς πολυμερής ή αν από την άλλη μεριά θα είναι υποχρεωτική η αλληλεγγύη, η επίδειξη αλληλεγγύης. Αυτό βέβαια θα εξαρτάται από τον τομέα και από το θέμα για το οποίο μιλάμε. Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλιστούν, να, να λαμβάνεται απόφαση για το ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά. Τρόποι συνεργασίας, μορφές αλληλεγγύης, ε, δράση συγκεκριμένων φορέων κλπ. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τον ρόλο των διεθνών παραγόντων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, ε, η Πατιαρμοστήρια της τους πρόσφυγες κλπ. Μέσω αυτών μπορεί να δείξει επίσης αλληλεγγύη. Θα πρέπει και αυτοί άλλωστε οι φορεί ε, να συμπεριλαμβάνονται στην αντισυσιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τι θα πρέπει να έχει υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ του δράσει. Πρώτον, οικονομικέ πτυχέ. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν γραμμές στον προπολογισμό για ε, προβλέψεις ε, ποσών για τα κράτη-μέλη, κονδυλίων προς τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στη διαχείριση των συνόρων τους. Επίσης, θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να δημιουργήσει συγκεκριμένα ταμεία. Πρέπει να ξαναδούμε αν τα μέσα τα οποία διαθέτουμε είναι επαρκή ή όχι. Πώς θα πρέπει να κατανέμονται και ποιους ε, στόχους θα πρέπει να έχουν στην αναθεώρηση της Frontex ίσως θα μπορούσαμε θα μπορούσατε να καλύψετε κάποιες αδυναμίες που έχουν εμφανιστεί και να λάβετε υπόψη για το θέμα της αλληλεγγύης. Και τέλος, θα μπορούσατε θα έπρεπε ενδεχομένως να εξασφαλίσετε ότι η αλληλεγγύη θα λαμβάνεται υπόψη και στην κοινοτική νομοθεσία. Κάθε φορά που υιοθετείτε ε, νομοθεσία, όπως ζητούμε την εφαρμογή της αρχής επικορικότητας, έτσι θα μπορούσατε να ζητάτε και την, και την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Συνεργασία. Άλλο γενικό συμπέρασμα, συνεργασία σε αυτά τα θέματα είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία ε, όχι μόνο ε, στους τομείς των συνόρων του ασύλου της μετανάστευσης αλλά και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η κατάρριξη των εσωτερικών συνόρων είναι μία από τις επιτυχίες μεγάλες επιτυχίες τη Ευρωπαϊκής Ένωση για τους πολίτες τη και για τι επιχειρήσεις. Το γράσο που διατηρεί αυτή το, μηχανισμό σε λειτουργία είναι η ικανότητα των κρατών μελών να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται το ένα το άλλο στη διαχείριση των συνόρων, στην, στην ε, αξιολόγηση του καθεστώτος ε, των, ε, των, και στην ένταξη των αλλοδαπών στις κοινωνίες τους. Συνεπώς, η αρχή της αλληλεγγύης του άρθρου 80 θα πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Βανχόιλε, και για την παρουσίαση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος εκκρεμούς θέματος αλληλεγγύης. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει αυτή την απουσία αλληλεγγύης, η οποία είναι απαράδεκτη. Όπου θεσπίζεται με την συνθήκη της Λισαβόνα το άρθρο 80, η υποχρέωση με την αρχή της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ήταν πηγή έπνευση αυτή η παρουσίαση. Αρχή η συζήτηση. Βλέπω ότι ο κύριος Μπουσούτιλ θέλει να κάνει πρώτος μια παρατήρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ξεκινώ ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, για τη μελέτη του, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θέλω να ευχαριστώ και τους συναδέλφους από, τις, ε, από το τμήμα των ιστορικών ε, πολιτικών, μελετών ιστορικών πολιτικών, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και το προέβλεψαν στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, Πρόεδρε, όπω είπατε, για εμά ω θεσμικό όργανο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν πάντοτε το όργανο το οποίο αγωνίστηκε για την ε, ε, ιδέα της ελληνικής. Αυτό δεν ε, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ελληνικής. Το γνωρίζουμε πολύ καλά τώρα πλέον. Πάνω απ' όλα όμως το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση. Εάν υπάρχει υπαρχής πολιτική βούληση, όπως είπε και ο μιλητής, πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ουσιαστικά να εκφραστεί και στην νομοθεσία για το άσυλο και στην νομοθεσία για τη μεταναστεύση, αλλά και στην υλοποίηση αυτών των νόμων η αλληλεγγύη, στις πολιτικές δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προχωρώ για να μιλήσω για τις θέσεις των άλλων θεσμικών οργάνων. Είναι σαφέστατα οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή. Είμαστε υπέρ του άρθρου 80, υπέρ της εφαρμογής του. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε την ίδια στάση από πλευρά Συμβουλίου. Με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να δυνατεί να συμφωνήσει σε μέτρα σχετικά με την αλληλεγγύη συμπεριλαμβανομένων και σε ορισμένε περιπτώσεις ε, θεμάτων σχετικών με την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, όπου, όπως είπε και ο εισηγητής, υπάρχει ακόμη ζήτημα ως προς την προσωρινή άρση εφαρμογής του κανονισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις. Προσέθεσε δε ότι υπάρχει δυνατότητα για αντισταθμιστικά μέτρα σε περίπτωση επανεγκατάστασης. Όμως κανένα από αυτά τα μέτρα, καμία από αυτές τις λύσεις δεν δέχεται να συζητήσει το Συμβούλιο και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η απουσία πολιτικής βούλησης. Για δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φρονώ ότι η Επιτροπή είναι πάντα στο πλευρό μας στην υπόθεση αυτή, στα θέματα της αλληλεγγύης και ότι εγώ θα ήθελα να δω πιο ε, θαραλέα πολιτική. Εάν δούμε το πακέτο για το άσυλο που έχει τεθεί επί Δεν υπάρχει καμιά θαραλέα νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα τη αλληλεγγύη. Υπάρχουν κάποιε πρωτοβουλίε, εκ των οποίων η μία αφορά και τη δική μου πατρίδα, τη Μάλτα. Αξιέπαινη πρωτοβουλία, αλλά πιστεύω πέραν αυτών θα πρέπει να προχωρήσουμε στην νομοθετική πρόταση που θα εδραιώνει την ε, αλληλεγγύη. Μία ερώτηση συγκεκριμένη για τον εισηγητή σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να διεκδικήσει κανεί ε, από τα δικαστήρια την επιβολή του άρθρου 80, σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να καταστεί καταναγκαστικό άρθρο αυτό ε, και να προβληθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, και αν ναι, με ποια κριτήρια, με ποια επιχειρήματα. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άρθρο της συνθήκης, το οποίο όμως δεν έχει εκφραστεί σε συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο ή δράσεις δε μάλλον. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορεί κανείς να επικαλεστεί το άρθρο αυτό για να προσβάλλει αυτή την απουσία δράσης, αυτή την παράληψη. Θα σταματήσω εδώ για να ακούσουμε και τους άλλους ομιλητές και ευχαριστώ και πάλι τον ομιλητή για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουσούτη, λέει ο πρόεδρος. Ο κυριος Παπανικολάου έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση. Και ευχαριστώ επίση και τον κύριο για τη συμφωνία μαζί του. Ε, με λίγα λόγια, είσαστε αισιόδοξο για το θέμα τη αλληλεγγύη. Θεωρείτε ότι οι όροι της ε, υλοποίηση αυτή θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στο θέμα αυτό. Και τι γνώμη έχετε για το ενδεχόμενο να μην μπορέσουμε να χειριστούμε το θέμα όπως το θέλουμε. Ευχαριστώ, Ιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και εγώ τον καθηγητή στην παρέμβασή του παρουσίασε ένα πλήρες οργανικό έγγραφο που θέτει φως ε, την αλληλεγγύη. Θεωρώ όμως ότι η αλληλεγγύη δυνάμει του άρθρου 80 και βάσει των άλλων διατάξεων της συνθήκης νομίζω ότι προβλέπεται επαρκώς. Η εφαρμογή λείπει. Δηλαδή, μεταξύ των προβλέψεων των νομοθετικών υπάρχει διαφορά και μεταξύ της συγκεκριμένη συμπεριφοράς και των συγκεκριμένων ε, εφαρμογών. Αναφέρεται επίσης και το θέμα της Frontex και η αναθεώρηση εντολής απαιτείται για τη Frontex για να γίνει αποδοτικότερη, πιο ευέλικτη, πιο κομψή και το θέμα αυτού και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών. 2014 θα έχουμε τις νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και θα υποστηρίξουν ε, πιστεύω και την διαχείριση των ε, συνόρων με μεγαλύτερη προσοχή στις συμφωνίες επανιστοχής που χρειάζονται που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρέμβασή του και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, ε, τη διεύθυνση αυτή που πρότεινε, ε, τη σημαντική αυτή μελέτη που είναι μια στιγμή που εμπλουτίζει τις γνώσεις ε, όλων μας και εκπονήθηκε από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ. Κυρία Βίξτρομ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ιβαν Χόιλε. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατη αυτή η δουλειά που έγινε και πραγματικά μας διευκολύνει ε, στην εξέταση του θέματος της μετανάστευσης και του ασύλου να μπορέσουμε να αναφερόμαστε, να παραπέμπουμε στη μελέτη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι πληρέστατη η έκθεση. Πραγματικά, κατά την άποψή μου, η αλληλεγγύη ακολουθεί δύο προσεγγίσεις. Είναι αφίδρομη η διαδικασία. Πρέπει όλοι να εφαρμόζουμε σωστά τους κανονισμούς. Και δεύτερον, όταν η πίεση επί ενός κράτους μέλους είναι μεγαλύτερη από ό,τι επί άλλων κρατών μελών, θα πρέπει τα άλλα κρατημέλη να βοηθάνε. Σωστά το λέει η έκθεση στα συμπεράσματά της, η εμπιστοσύνη είναι βασικό θέμα. Όταν ήρθαν τα εσωτερικά σύνορα, όπως έγινε, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Να θεωρούμε δηλαδή ότι γίνεται σωστή χρήση έλεγχος των εξωτερικών σύνορων και πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Όμως χρειάζεται μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης για να εξασφαλίζεται η αλληλεγγύη, χρειάζεται και πίστη για να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη. Αλλά για να εξασφαλίζεται αυτή η πίστη χρειάζεται αλληλεγγύη. Και έχουμε έναν κύκλο ο οποίος αποτελεί και τη βάση της Ευρωπαϊκής Ενώσης και είναι καλός κύκλος αυτός, όχι μόνο όσον αφορά τη μετανάστευση, αλλά εν γέννη. Κατά την άποψή μου είναι ξεκάθαρο ότι όλοι ωφελούνται αν ο κύκλος αυτός είναι σταθερός, αν υπάρχει μια πολύ στερή βάση εμπιστοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι δεν χρειάζεται και πολύ για να καταστραφεί και να διαλυθεί ο μηχανισμός. Όταν η Ιταλία δίνει άδεια για ελεύθερη μετακίνηση των τυνησίων μεταναστών, χάνει την εμπιστοσύνη η Ιταλία από τα άλλα όπως η Γαλλία χάνει την εμπιστοσύνη στην Ιταλία. Και χωρίς εμπιστοσύνη η Γαλλία πιθανότατα δεν θα δείξει αλληλεγγύη και δεν θα βοηθήσει την Ιταλία να χειριστεί την εισρωή των μεταναστών. Και όταν η Δανία θέλει να επαναφέρει τους μεθοριακούς ελέγχους, δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τα άλλα κράτη-μέλη και γι' αυτό δεν θα δείξει την παραμικρή αλληλεγγύη. Ξαντάλλαγμα, η Δανία θα πρέπει να αναμένει ότι και τα άλλα κράτη-μέλη δεν θα είναι πιστά έναντι αυτής οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται για να αυξήσουμε την πίστη, την αλληλεγγύη θα ενισχύουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πάντα θα υποστηρίζω τέτοια μέτρα. Σας παρακαλώ όμως πείτε μας πώς εμείς σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι αυτός ο κύκλος της εμπιστοσύνης και πίστης και αλληλεγγύης ε, θα οικοδομηθεί. Από πού ξεκινάμε την κατασκευή του κύκλου. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ένας τομέας, ένας χώρος εμπιστοσύνης. Προσπαθούμε, αλλά δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ, η κυρία Φλότ έχει το λόγο τώρα. Είναι αλήθεια. Ε, είναι εντυπωσιακό ε, να ακούμε μια μελέτη για την αλληλεγγύη, γιατί στην σημερινή επικαιρότητα βλέποντας τι γίνεται στο άσυλο, την μετανάστευση και τα εξωτερικά σύνορα, ε, κανείς ε, αντιλαμβάνεται ότι για να μιλήσει για αλληλεγγύη πια πρέπει να είναι ακραίος ακτιβιστής ε, ε, ε, ή υπέρ της Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Και αυτό είναι το πρόβλημα της αλληλεγγύης. Γιατί δεν υπάρχει αλληλεγγύη χωρίς απόδειξη αλληλεγγύης, όπως δεν υπάρχει και έρωτας χωρίς απόδειξη αυτού του έρωτα. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καθόλου αλληλεγγύη. Δυστυχώ. Τώρα, σε αυτή την ιδέα, ή ε, σε αυτό το, το, κεφάλαιο, ε, κάποιοι θεωρούν ότι η αλληλεγγύη είναι ένα βάρος που θα πρέπει να το μοιραστούμε. Αυτό γίνεται όλο και λιγότερο σωστό και δίκαιο για τη μετανάστευση. Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εργασίε που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη για την ανάπτυξη μια θετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί οι μετανάστες ε, σε λίγο θα ενδεχομένως θα γίνουν ε, αντικείμενο έρηδας ανάμεσα στα κράτη-μέλη για το ποιος θα, τα, τους ε, υποδεχτεί πρώτος. Συνεπώς αυτή η αλληλεγγύη δεν είναι ένα άχθος πλέον. Θα πρέπει να τη δούμε διαφορετικά. Οι συμφωνίες του Δουβλίνου, για παράδειγμα, ε, δεν είναι αλληλέγγυες. Όσο και, εμείς, όσο και αν ε, καλούμε εμείς ε, για την, απόδειξη, στην επίδειξη αλληλεγγύης. διότι οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν συγκεκριμένες ευθύνες για συγκεκριμένα κράτη. Οπότε ε, μέχρι τώρα είναι στη διακριτική αυχαίρεια του κάθε κράτους μέλους να δείξει η αλληλεγγύη ή όχι. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η αλληλεγγύη είναι, υπέρ, είναι κοινό, υπέρ του κοινού συμφέροντος. Μόνο έτσι θα ανοίξουμε ένα ρήγμα στη σημερινή κατάσταση. Αν δεν το δούμε έτσι, πολύ δύσκολα θα εφαρμόσουμε στην πράξη δράσεις αλληλεγγύης. Συνεπώς και την ίδια την έννοια της αλληλεγγύης. Η κυρία Έρνστ έχει το λόγο. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα με την αλληλεγγύη. Όποιος ε, φωνάζει πιο δυνατά έχει και περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι ως Γερμανίδα βουλευτής μου φαίνεται λίγο δύσκολο να αιτιολογώ την κατάσταση την, ε, μάλλον την αρχή της ελληνικής δεν της Ιταλίας. Αντιλαμβάνομαι ποια είναι η κατάσταση μεν, αλλά μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία στην περίοδο του 90, δεκαετία του 90, ήρθαν 300.000 πρόσφυγε από την πρώην Ιουκοσλαβία. Και του υποδεχθήκαμε εμεί στη Γερμανία, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, δεν κλείσαμε σύνορα. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε κάπω πιο θεμελιώδη ζητήματα στην αλληλεγγύη. βεβαίω, βεβαίω αλληλεγγύη, και για όνομα του Θεού δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τη βασική αρχή τη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί εδώ. Αλλά Εάν δεν συστούμε το Δουβλίνο 2, εάν αφήνουμε τα πράγματα όπως έχουν, εάν δεν, δεν εξασφαλίζουμε μια ουσιαστική αλλαγή, όσο και να μιλάμε, τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θα έρχονται οι μετανάστες και θα επιβαρύνουν συγκεκριμένα κράτη, τα κράτη στα οποία έχουν αφιχθεί κυρίως. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε πρακτικές και ε, ικανοποιητικές λύσεις στο θέμα της αλληλεγγύης. Επίσης σημαντική είναι η πρότασή σας, η προτάσή σας μάλλον για την προστασία των ετούντων του άσυλου. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφοροποιημένη θεώρηση του ετούντος ή της ετούντος του άσυλο που έρχονται στις χώρες μας προερχόμενοι από τις χώρες Αφρικής. Καταρχάς δεν ζητούν το άσυλο. Πρόκειται κυρίως για αλλοδαπούς μετανάστες που είχαν εργαστεί στη Λιβύη πλήστον, από την Ιγυρία, από άλλα κράτη, ως γκάσταρμπάιτερ δηλαδή και τώρα έρχονται πάλι στις χώρες μας για να αναζητήσουν μια νέα θέση εργασίας. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, το ξέρουν πολύ καλά ε, δεν μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους, γιατί αυτή είναι η ουσία, και ως εκ τούτου ζητούν κάποια λύση και πρέπει και εμείς να βρούμε λύση για τους ανθρώπους αυτούς. Φερειπίνη προσωρινή προστασία, όπως και εσείς πιστεύω υπενεχθήκατε. Λύσεις τις οποίες, ε, οι οποίες θα μας επέτρεπαν να τους προσφέρουμε για ένα χρονικό διάστημα μια λύση, μια θέση εργασίας και που ταυτόχρονα θα τους διευκόλυναν και να ε, επιστρέψουν στις χώρες τους αργότερα, αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα είμαστε αλληλέγγυοι και σε συνεργασία και με εκείνους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο φόρτο να ε, υποδεχθούν, που φτάνουν μέχρι τις 700.000 ε, μεταναστών στα σύνορά τους. Και επίσης την αλληλεγγύη θα ήθελα να την συστήσουμε και ως προς την ε, επανεγκατάσταση, resettlement, διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ε, χωρίς να αναλλάξουμε στάση στην υπόθεση αυτή. Τι σημαίνει εκούσια επανεγκατάσταση. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες θα λειτουργούν ε, κατά τρόπο εκούσιο εθελοντικό, αλλά ταυτόχρονα ίσως θα πρέπει να διαρωτηθούμε μήπως χρειάζεται και να επιβάλλουμε την υπο... ή να αναγνωρίσουμε μάλλον την υποχρέωση στην αρχή αυτή της επανεγκατάστασης ως έννοια της αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι σε μια σειρά θεμάτων ε, μπορούμε να προτείνουμε τροποποιήσεις, αλλαγές οι οποίες θα σημάνουν και ουσιαστική εφαρμογή της αλληλεγγύης, ώστε να μην παραμένει αυτή γράμμα κενό. Και να βοηθάει τελικά στην επίλυση των προβλημάτων, εκείνων που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εάν δεν έχει κάνει άλλα σχόλια, εάν δεν σηκώνει κάνει το χέρι του, α δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Βαν Χούιλε για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ για τι πολύ αυστοχές παρατηρήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση σα, για το δυναμικό, για τις ικανότητες. Δεν έχει απαντηθεί ακόμη το ζήτημα αυτό. Το μόνο που μπορούμε να, ε, με το οποίο μπορούμε να το συγκρίνουμε είναι η αρχή της αλληλεγγύης και της ε, συνεργασίας συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αν κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριστεί το δικαστήριο την αρχή αυτή και στο σε ποιο βαθμό την έχει θεωρήσει αναγκαστικού δικαίου, βλέπουμε ότι δεν θεωρεί πω έχει άμεση ισχύ η διάταξη αυτή. Αντίστοιχα σε άλλε περιπτώσει, ότι δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε ε, προσφυγή για παραβίαση, σε συνδυασμό όμω με άλλα καθήκοντα τα οποία έχουν εντωμεταξύ ενσωματωθεί μέσα στο πλέγμα το νομοθετικό του ευρωπαϊκού δικαίου. Άρα, εάν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, η πιθανή απάντηση που θα μπορούσα να δώσω χωρίς όμως να μπορώ να προβλέψω τι είδους νομολογία θα προκύψει από το δικαστήριο σε μια ενδεχομητική υπόθεση θα ήταν ότι θεωρώ μάλλον δύσκολο δυνάμει του άρθρου 80 και μόνο να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση ε, με το επιχείρημα ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 80. Θα είναι μάλλον δύσκολο να κερδίσει μια τέτοια υπόθεση. Αυτή ήταν και μια από τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί στα προπαρασκευαστικές εργασίες ε, της ε, ε, για τα ευρωπαϊκά όργανα όπου είχε επισημανθεί από κάποιον από τους μετέχοντες ότι θα είναι πρόβλημα η ιδέα της ε, επίκληση στο δικαστήριο για άμεση εφαρμογή αυτού του άρθρου της αλληλεγγύης γιατί δεν ήταν σαφέ με τι είδου κριτήρια θα μπορούσε να γίνει η επίκληση και τι είδου νομικέ διαδικασίε, οι δικαστικές διαδικασίες θα μπορούσαν να τεθούν σε ε, λειτουργία δυνάμει αυτού του άρθρου. Αυτή είναι η κατάσταση πάντω μέχρι τώρα, δεν είναι πολύ σαφή όπω σα λέγω. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί το άρθρο αυτό, το 80 δηλαδή, αυτόνομο και μεμονωμένο να να τύχει επικλήσεως ενώπιον δικαστηρίου και να οδηγεί σε νομικές συνέπειες. Πάντως ένα σημαντικό θέμα είναι μια απόφαση, είναι μια διάταξη που ισχύει και έχουμε δει πολλές φορές ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έχει λάβει αξιόλογες και εντυπωσιακέ αποφάσεις σχέση με κάποια άρθρα των συνθήκων. Πάντως θα πρέπει να επισημάνω ότι είμαστε ακόμα σε μια εμβριακή φάση ως προς την αρχή της αλληλεγγύης και ίσως χρειαστεί ακόμη περαιτέρω επεξεργασία και ανάπτυξη. Αυτό ήταν το δικό μου σχόλιο. Για τον κύριο Παπα-Νικολάου ερώτηση και παρατήρηση αισιοδοξία προ τα ζητήματα της, της αλληλεγγύης, βραχυπρόθεσμα, προβλέψεις. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις από τις συνεντεύξει που έχουμε διεξαγάγει και έχουμε διεξαγάγει συνεντεύξει με εκπροσώπους από τα ευρωπαϊκά όργανα, τι διεθνεί Οργανώσει, τα κράτη-μέλη και τα όμορα, μάλλον και τα κράτη που έχουν εξωτερικά σύνορα και τα εσωτερικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων σε αυτό το πεδίο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συνείδηση του προβλήματος, ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει δηλαδή ευρωπαϊκή πολιτική. Εάν θέλουμε η Ευρώπη να λειτουργεί χωρίς εσωτερικά σύνορα, θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών σύνορων. Κάποιοι προβάλλουν το επιχείρημα ε, ότι οι συνοριοφύλακες πλέον δεν εργάζονται για να προστατεύσουν μόνο τα δικά τους σύνορα, αλλά ότι προστατεύουν συνολικά τα σύνορα της Ευρώπης. Και αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και μια αφύπνιση, μια ευαισθητοποίηση ως προς το πανευρωπαϊκό του έργου τους. Σε αυτό μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξη. Ίσως υπάρχει κάποια ελπίδα να δούμε πρόοδο στη συνείδηση του θέματος αυτού. Το βλέπουμε σε κάποιες από τις συνεντεύξεις που έχουμε δεξαγάγει. Και υπάρχει εξέλιξη όπως λέγω. Πρόβλημα βλέπω όμως εκεί όπου στη δεύτερη φάση αυτή της διαδικασίας, είτε πρόκειται για την νόμιμη μετανάστευση, είτε πρόκειται για το άσυλο, έχουμε να συνδυάσουμε αυτή την ιδέα με τις συνέπειες νομικές. Δηλαδή εκεί που γίνεται λόγος για διαχείριση συνόρων και φύλαξη συνόρων δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όταν πια τίθεται και το ερώτημα της νόμιμης μετανάστευσης, του ασύλου, των προσφύγων, τότε πια τα πράγματα μπερδεύονται και δυσκολεύουν διότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κανείς έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μακροπρόθεσμη διάρκεια και είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλήξουμε συμφωνία σε συνεννόηση για το ποιο θα αναλάβει τι και ποιον. Άρα η πανευρωπαϊκή ενδεχομένως ιδέα της συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί αν αυτό ακριβώς με ρωτούσατε. Δεν έχει δηλαδή υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση ότι κανεί φυλάσσει τα σύνορα ολόκληρης της και δεν νομίζω ότι, γρήγορα, θα το δούμε αυτό γρήγορα. Για την ε, νόμιμη ή παράτυπη μετανάστευση βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις ε, δηλαδή στην ε, νόμιμη, ή στην ε, σύνομη μετανάστευση κάποιοι δίνουν απαντήσεις μάλλον εντυπωσιακές, αναπάντεχες. Πολλές φορές βλέπουμε θετική ε, στάση απέναντι στην ιδέα της ε, μετανάστευσης, την οποία ε, στάση θα μπορούσαμε περαιτέρω επεξεργαζόμενοι να ενισχύσουμε, να διαδώσουμε και να βελτιώσουμε την αποδοχή της σύνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα τώρα να φτάσω στο ερώτημα που ακούστηκε νωρίτερα ως προς το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι ρόλο μπορεί να διδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μπορεί να διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κάνω διάκριση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων. Οι βραχυπρόθεσμες, όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι η δυνατότητα φερειπίν του να επανεξεταστεί η Frontex, η χρηματοδότησή της ή να ανοίξει μια συζήτηση επί του προϋπολογισμού της, όπου μπορεί να διδραματίσει σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο και να έχει με τις αποφάσεις του άμεσο αντίκτυπο στις χώρες μέλη ή στην επιβάρυνση που επομίζονται ε, αυτές, δηλαδή με άμεσο αντίκτυπο. Και υπάρχει και η μακροπρόθεσμη θεώρηση, λίγο πολύ αυτό το οποίο έθεσε με τις παρατηρήσεις κυρία Έρνστ, ότι δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι μια γενική συζήτηση, ένας διάλογος για το πού θέλουμε να, ε, τι, στόχο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε με τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το θεωρούμε ότι η μετανάστευση, το άσυλο, η διαχείριση των συνόρων είναι η πραγματική, η γνήσια οδός για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρώπης, θα πρέπει ταυτόχρονα κάπως να ορίσουμε αυτή την έννοια της μετανάστευσης, όπου εντοπίζεται και ο, η αντίφαση μεταξύ των όσων μπορεί να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής δηλαδή, και των όσων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως μια ευρεία ιδέα της μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή πλαίσια. Μιλισμονούμε ότι σε 20 χρόνια, με δεδομένε δημογραφικέ εξελίξει που σημειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστούμε πολύ νέο αίμα και ω εκ τούτου έχουμε ευθύνε. Έχουμε ευθύνε όμως και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τους ε, πρόσφυγες, για κάθε άλλον που είναι ε, σε ανάγκη προστασίας, που, έχει, ε, που χρήζει προστασίας, όπως σε παραδείγματα θύματα των ε, λαθρεμπόρων ανθρωπίνων όντων. Όλα αυτά τα πράγματα στα οποία θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα και επίση θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα σε σχέση με το Συμβούλιο, διότι εκεί εκφράζονται εθνικέ αντιδράσει, εθνικέ αντιδράσει οι οποίε ουσιαστικά τείνουν προ την αντίθετη κατεύθυνση της, ε, σε σχέση με τη δημιουργία ε, ενό ευρωπαϊκού χώρου. Μα λένε δηλαδή ότι α εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να πουληθεί εντό εισαγωγικών αυτή η ιδέα, δεν πουλιέται, δεν μπορούμε να την προβάλλουμε, πρέπει να έχουμε πιο προστατευτική στάση έναντι τη μετανάστευση ή ε, εξελίξεις άλλωστε που είδαμε τους τελευταίους μήνες είναι ξεκάθαρες. Επιβαρύνεται ε, με ε, αφήξεις μεταναστών μία χώρα και η άλλη χώρα κλείνει τα σύνορά της και δεν συνεργάζεται. Άρα είναι σαφέ ότι μπορεί μια κοινοβουλευτική συνέλευση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να γίνει συζήτηση πιστεύω στο δικό σα επίπεδο για το τι επιδιώκουμε με τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί όμω να έχουμε τη θεώρηση, την εθνική, μόνο το εθνικό πρίσμα, αλλά, τον τρόπο με τον, αλλά να αναζητούμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε η μετανάστευση να καταστεί δυνατή ε, σε βαθμό που είναι σύνομη και χωρί εσωτερικά σύνορα. Αυτό μέσα σε μια πολιτική που και θα χαράσει την ε, νομοθεσία και θα αφήνει ανοιχτό το πεδίο για το δημόσιο διάλογο, όπως έχουμε δει και σε, άλλα, σε άλλους τομείς, σε άλλα θέματα, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητά Βανχόλε για αυτή την ε, μελέτη σημείο αναφοράς προς περαιτέρω συζήτηση. Ε, λοιπόν, για να δώσουμε περιεχόμενο στην αλληλεγγύη, για να έχει νόημα. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτά για την ώρα, σαν αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Η Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ, ήδη κατέφθασε. Περιμένει να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011. Ευχαριστώ καθηγητά και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Λοιπόν, προσέξτε, την προσοχή σας παρακαλώ συναδελφοί. Καλωσορίζουμε εκ νέου στην Επιτροπή, στην αίθουσα της Επιτροπής Ελευθεριών, την Επίτροπο Μάλστρομ για δεύτερη φορά σήμερα. Την ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ έτοιμη να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 και την προετοιμασία του προγράμματος εργασιών του 2012. Να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων εφαρμόζει ουσιαστικά υλοποιεί τη Συμφωνία Πλαίσιο όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε να ακούσουμε τι γίνεται με τις, προτεραιο... τις προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για φέτος. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Επίτροπος και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Κυρία Επίτροπε, κυρία Μάνστρομ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ναι, στον τομέα μου τα πάντα είναι ήρεμα, δεν υπάρχουν ε, προβλήματα. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποια ζωή στο θέμα για να μην αποκοιμηθείτε κιόλα. Βέβαια, όπως πάντα, είναι χαρά μου που είμαι εδώ για να παρουσιάσω κάποιες πρωτοβουλίες και να σε ενημερώσω για τις εξελίξεις. Και με τα χαράς να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η κατάσταση στη Νότια Μεσόγειο κυριάρχησε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη δική σας δουλειά, στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο δικό μου προσωπικό πρόγραμμα. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσω, αναφερόμενη στην ανακοίνωση για τη μετανάστευση που παρουσίασα πριν από 10 μέρες και υπό το φως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου που θα έχει στο επίκεντρο βασικό θέμα τη μετανάστευση και θα συζητηθούν πολλά από αυτά τα ζητήματα. Η ανακοίνωση όσον αφορά τα μεταναστευτικά ζητήματα προσπάθησε να καλύψει τη γενική εικόνα, τη συνολική εικόνα της μετανάστευσης. Εκάλυψε τα πάντα από μετανάστευση, νόμιμη μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, ε, πολιτική ασύλου, έλεγχη συνόρων, Frontex, θεωρήσεις, Schengen κλπ. Ε, για να προσπαθήσουμε να απομακρυνθούμε λίγο από τη συζήτηση που διεξήχθη με θέμα της εξελίξης στην Ανατολ... στη Μέση Ανατολή Όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική ασύλου και να δίνουμε προστασία σε εκείνους που ζητούν διεθνή προστασία αν δεν έχουμε πολιτική ασύλου η οποία να είναι συνεκτική και αν δεν έχουμε αποτελεσματική νόμιμη ε, μετανάστευση αν δεν έχουμε συστήματα ένταξης, δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε πολιτική θεωρήσεων που είναι αξιόπιστη και αν δεν έχουμε μεθοριακούς ελέγχους και αν δεν έχουμε μια πολιτική για να αντιμετωπίσουμε την παράτη μετανάστευση δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν δεν έχουμε επιτρο... μια πολιτική επιστροφών, επανεισδοχής που να είναι ανθρώπινη. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα από όλα αυτά αν δεν συνεργαστούμε με τρίτες χώρες, αν δεν συνεργαστούμε με πιο συντονισμένο τρόπο ε, από ό,τι κάναμε κατά το παρελθόν. Θα ξεκινήσω με το θέμα του Σέγγεν, διότι αυτό δημιούργησε πολλές συζητήσεις, πολλά ερωτηματικά και θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα ο πρόεδρος Μπαρόσο και εγώ στην Ολομέλεια πιο πριν στο μήνα ότι δημιουργία του χώρου Σέγγεν χωρί εσωτερικά σύνορα και χωρί εσωτερικού ελέγχου είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είναι ένα δώρο προ του Ευρωπαίου πολίτε και θα προασπιστούμε αυτό το δώρο. Είναι ένα ισχυρό σύμβολο τη ευρωπαϊκή ολοκληρώσεω που δεν χρειάζεται να δείξουμε το διαβατήριο πηγαίνοντα με αυτοκίνητο από τη Φιλανδία στην Πορτογαλία ή από τη Μάλτα στην Εστονία. Πρέπει να πάρετε το φέρι βέβαια. Τέλο είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό και θα πρέπει να το προστατεύσουμε και να το προωθήσουμε. Και καλωσορίζω το ότι υπερασπιστήκατε στεναρά εσείς στο Σέγκερ και ότι έτυχα υποστήριξεω του Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, όχι μόνο τα πρόσφατα, αλλά και πριν από αυτό, το σύστημα δεν είναι τέλειο και η αξιολόγηση του Σέγγεν μέχρι τώρα κοίταζε μόνο προς τα πίσω, προς το παρελθόν. Θα θυμόσαστε ότι πέρσι τον Νοέμβριο παρουσίασα μια πρόταση ούτω ώστε να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, να γίνεται καλύτερη διαχείριση του Σέγγεν μέσω καλύτερου μηχανισμού αξιολογήσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχοντας έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, διαφορετικά από σήμερα που τα κράτη-μέλη αυτοαξιολογούνται. Επίσης, το χρειαζόμαστε αυτό, ούτω ώστε να ανοίξουμε, να διευκολύνουμε την κατάσταση για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να μπουν στο Σέγγεν πρέπει, πληρούν τα κριτήρια τα τεχνικά, αλλά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη από τα άλλα κράτη-μέλη. Χρειάζεται εργαλεία να αντιδρούμε και να μπορούν τα κράτη-μέλη να χειρίζονται αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χρειάζεται ενίσχυση του ελέγχου, τη παρακολουθήσεω και πρέπει να εντοπίσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη θέση μα, ούτω ώστε να βοηθούμε ένα κράτο μέλο αμέσω όταν αυτό το κράτο μέλο ε, δέχεται πάρα πολλέ μεγάλες πιέσει ή για τον ένα τον άλλο λόγο δεν μπορεί να ελέγξει τα σύνορα Έχουμε βοηθήσει με τη διαδικασία, με την επιχείρηση Rabbit την Ελλάδα και έχουμε όλα τα εργαλεία και πρέπει να έχουμε όλα τα εργαλεία πολύ έγκαιρα να βοηθάμε τα κάτι μέλη και θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα για να έχουμε συστάσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά ε, με το πώς τα άθρα του κεκτημένου του Σέγγεν θα πρέπει να ερμηνεύονται. Τώρα γενικότερο στόχος είναι να εντοπίσουμε πιο νωρί τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις ταχύτερα δυνατόν, να ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο να επανεισαχθούν μέτρα για ελέγχου εσωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να γίνεται αυτή η προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντοπισμό των προβλημάτων και όταν το κάνουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο λιγότερε οι πιθανότητε να επανεισαχθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Υπάρχουν εξαιρετικέ περιστάσει βέβαια, όπου ίσω οι έλεγχοι στα σύνορα μπορούν να, θεσ... να επαναφερθούν προσωρινά. Προβλέπεται στη συνθήκη για μεγάλε αθλητικέ εκδηλώσει ή τρομοκρατικέ απειλέ, οι επιθέσει προβλέπεται και έγινε αυτό. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πάντα τα κάτι μέλη πολύ προσωρινά να κάνουν ελέγχους, να δημιουργούν ελέγχους στα σύνορα σε κατεπίγουσες καταστάσεις, σε περιπτώσεις ανάγκης. Προτίθεται να κάνει πριν τι διακοπέ του καλοκαιριού Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσει για να βελτιώσουμε το μηχανισμό αξιολόγηση ελέγχου, την ευρωπαϊκή διάσταση επίση τη διακυβέρνηση και αυτό θα επιτρέψει με την υποστήριξή σα να καλύψουμε κάποια από τα κενά που έχουμε τώρα, να έχουμε ένα πιο ισχυρό σύστημα στο μέλλον. Επίση, έγινε συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για την Νότια Μεσόγειο και όπως είπα επανειλημμένα, όταν αναφέρθηκα στις διάφορες δράσεις που αναλάβαμε ε, όσον αφορά αυτό το θέμα, σήμερα το πρωί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε κάποια μέτρα σχετικά με το ζήτημα αυτό, ε, μια ανακοίνωση «Διάλογος, η κινητικότητα, μετανάστευση και ασφάλεια για την Νότια Μεσόγεια». Προτείνουμε ένα μοντέλο για περαιτέρω επαφές με αυτές τις χώρες, ξεκινώντας από την Τινησία, την Αίγυπτο και το Μαρόκο να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για συνεργασία για κινητικότητα με ένα ευρύτατο φάσμα σημείων. Θέματα ασφαλείας συνόρων, σύστημα ασύλου, μετανάστευση, διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης και πώς να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα για τις θεωρήσεις, για τη διευκόλυνση χορηγήσεως θεωρήσεων και υπό κάποιους όρους βεβαίως, κάποιες συνθήκες, πιο μακροπρόθεσμα να καταβάλουμε προσπάθειες για περαιτέρω απελευθέρωση, χαλάρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι υποφελέ και για εκείνου και για μας και αυτό αποτελεί ένα τμήμα τη γενική προσεγγίσεω όσον αφορά τη μετανάστευση. Οθετήσαμε επίση τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο, το σύμφωνο αν θέλετε που η Γαλλική Προεδρία του 2008 δημιούργησε. Αυτή η έκθεση είναι άκρο τεχνική, αλλά συνοψίζει πολύ καλά τι έγινε και τι πρέπει να γίνει ακόμα στα κράτη-μέλη. Επίσης, υιοθετήσαμε ένα σχέδιο κανονισμού όσον αφορά τις απαιτήσει για χορήγηση θεωρήσεων μετά από την έγκριση του κανονισμού για τη θεώρηση. Επανειλημμένα έχει τροποποιηθεί ο σχετικός κανονισμός και η πρόσφατη τροποποίηση εστιάστηκε στις θετικούς και αρνητικούς καταλόγους που έχουν προσαρτηθεί στον κανονισμό. Ξέρετε πόσο σημαντικέ είναι αυτέ οι εξαιρεσει για μένα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι από τα πιο καλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να κάνουμε τον κόσμο να πλησιάσει ένα τον άλλον και να δημιουργήσουμε ε, περισσότερες για τι επιχειρήσει, Θα το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε και με τα Δυτικά Βαλκάνια και με άλλε χώρε. Είδαμε όμω ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά καταχρήσει σε κάποια κράτη-μέλη και σήμερα αν απομένουν προβλήματα για την, ε, που ίσως οδηγούν σε θέσπιση εκ νέου τη θεωρήσεω οφείλεται σε αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται μια ρήτρα διαφύλαξη που θα χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικέ περιστάσει και ελπίζω να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Πρέπει να υπάρχει για την προστασία τη ακαιρεότητα του συστήματο. Και να μα εξασφαλίζει ότι θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μέσω προγραμμάτων ε, από υποχρέωση θεωρήσεω με άλλε χώρε. Θα έχουμε ένα άρθρο διαφύλαξη, αν θέλετε, ρήτρα διαφύλαξη. υπό εξαιρετικέ περιστάσει, έσχατο μέτρο δεν αφορά καμία περιοχή του κόσμου, καμία συγκεκριμένη χώρα, δεν χρησιμοποιηθεί ε, κατά ιασδήποτε χώρα, όπως με ρώτησε ο σήμερα, εκπρόσωποι του τύπου, θα είναι απλώς μία ε, ρήτρα διασφάλισης. Έσχα το μέτρο αν υπάρχουν ε, περιπτώσεις παραβιάσεων κλπ. Και παράλληλα με όλα αυτά, χρειάζεται βέβαια να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για το θέμα των της μετανάστευσης, ε, νόμις μετανάστευσης, εποχιακούς εργαζόμενους, ενιαία άδεια ε, και μετα, μετακινήσεις στο ιστορικό μιας εταιρείας. Μετά, το πακέτο άσυλο. Πακέτο ασύλου. Για να ολοκληρώσουμε τις ε, πρωταβουλίες μας και να προετοιμάσουμε το, συμβόλιο Κορφής του Ιουνίου, η τροποποιημένη πρόταση για την ε, οδηγία ασύλου και η, ε, οδηγία, η επιτροπημένη οδηγία για τους όρους υποδοχής θα είναι έτοιμες ε, στις αρχές Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα των κρατών μελών, τροποποίησαμε λίγο τις προτάσεις μας χωρίς να μειώσουμε τη φιλοδοξία μας. Ελπίζω ότι με τη βοήθειά σας τον Ιούνιο θα τα καταφέρουμε να κλείσουμε το θέμα φτάνουμε κοντά στο 2012 και θα πρέπει να βιαστούμε. Η Κομισιόν επίσης εργάζεται και στο θέμα της ένταξης, άλλο σημείο κλειδί της μετανάστευσης. Ε, το φόρουμ της ε, ένταξης ε, το φιλοξενήσαμε χτες, δηλαδή και η ΟΚΕ. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλους τους τοπικούς παραγόντες γιατί η ένταξη γίνεται σε τοπικό επίπεδο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και με αυτόν τον τρόπο θα ε, εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τους μηχανισμούς και τους δείκτες που φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα και θα υιοθετήσουμε μια ανακοίνωση πριν το καλοκαίρι. Όχι νομοθετική πρόταση, μια ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής. Για το θέμα των καταστάσεων στοιχείων επιβατών έχουμε προχωρήσει διαπραγματεύσει με την Αυστραλία. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά όταν σχηματιστεί η κυβέρνηση εκεί και προχωράμε γρήγορα και στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Ενημέρωσα τους συντονιστές για αυτό το ζήτημα. Το θέμα του πακέτου τώρα των ευφυών συνόρων είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ή δυνατόν πριν το καλοκαίρι. Ε, περιλαμβάνει το σύστημα εισόδου-εξόδου και ε, ε καταγραφής των, ε, των εισερχομένων. Θα οδηγήσει αυτό το σύστημα σε μια καινούργια γενιά συνοριακών ελέγχων που θα βασίζεται σε καινούργια τεχνολογία. Όμως, απαιτεί σημαντικέ επενδύσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών, τη πληροφορία ε, ψηλού και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα και την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα προγράμματα, τεχνολογικά προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν πιλωτικά και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα ακούγοντας τους ενδιαφερόμενους, διαβάζοντας τις μελέτες ε, αντικτύπου κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο και με εσάς και με το Συμβούλιο πριν υποβάλουμε νομοθετική πρόταση. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι τα τρία όργανα, θεσμικά όργανα θα συνεργαστούν γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλα project ε, και οικονομικά αλλά και γενικότερα το βελνικές τους είναι ε, πολύ πλατή. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας εργασίας με τα μέλη σας, ενδεχομένως κοιτάω τον κύριο Κοέλιο αλλά και τους υπόλοιπους ε, για να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Επίσης να σας ενημερώσω και τελειώνω για την πρόοδο της ανάπτυξης ενός συστήματος παρομοίου με το TFTP. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους φορείς, Europol, κράτη-μέλη, SWIFT κλπ. Ε, για να το συζητήσουμε. Από τις συζητήσεις προέκυψε, προέκυψαν τρία σενάρια. Πρώτον, ένα κεντρικό σύστημα. Δεύτερον, ένα αποκεντρω... Ε, μάλλον ε, ένας αριθμός αποκεντρωμένων συστημάτων ή ένα μεικτό σύστημα. Η συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες οδηγεί περισσότερο προς το ανάμεικτο σύστημα. Το μεικτό σύστημα. Είναι τεχνικά περίπλοκο, Συνεπώ θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία δύο σταδίων. Τον Ιούλιο θα παρουσιάσουμε τις διάφορες ανακτικέ λύσει, τα διάφορα σενάρια και θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί σας και με το Συμβούλιο πριν υποβάλουμε συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα γιατί είναι ευαίσθητο. Τώρα, προστατεύοντα την ε, νόμιμη οικονομία. Είναι προτεραιότητά μα όχι μόνο για τη στρατηγική 2020, αλλά και, για, γιατί είναι ένα σημαντικό ε, τρόπο να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Από την αρχή τη θητεία μου είχα πει ότι θα αποτελέσει μία από τι προτεραιότητε μου, όπω και η ε, διάσταση τη ασφάλεια. Τι επόμενε εβδομάδε θα υποβάλουμε πρόταση. Σε μερικέ εβδομάδε λοιπόν θα διαθέτετε, θα έχετε στο τραπέζι σας ένα πακέτο εναντίον της διαφθοράς και από τη βάση αυτού η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια ανακοίνωση ε, που θα προβλέπει και τακτική αξιολόγηση των προσπαθειών των κρατών μελών να καταπολεμήσουν το, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε για να πετύχουμε το, ρόλο, το, το, στόχο της μείωσης της διαφθοράς. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει την προθυμία να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το πακέτο και ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί σύντομα. Θα προτείνουμε επίσης ένα καινούριο νομικό πλαίσιο για την κατάσχεση και ανάκτηση ε, των ε, παρανόμων ε, εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την αξιολόγηση της ε, ε, εφαρμογής της οδηγίας για την διατήρηση δεδομένων. 22 κράτη-μέλη την έχουν εφαρμόσει, Γερμανία, Ρουμανία και Τσεχική Δημοκρατία όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα συνταγματικά με το συνταγματικό του δικαστήριο η αξιολόγηση δείχνει ότι δεν έχει εναρμονιστεί η οδηγία με, με εναρμονισμένο τρόπο, με ενιαίο τρόπο. Ε, η οδηγία προβλέπει το πώς ε, αποθηκεύονται τα στοιχεία, ποιος ε, έχει πρόσβαση σε αυτά και για ποιους λόγους, αλλά δίνει πολύ ελευθερία στα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν κατά το δοκούν, οπότε ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η έκθεση εντοπίζει τα διδάγματα των τελευταίων πέντε ετών. Είναι διδάγματα ε, τα οποία μας ε, δείχνουν ότι τόσο οι επιχειρήσει όσο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια. Θα αρχίσουμε λοιπόν να, προετοιμάσουμε, να προετοιμάζουμε την αναθεωρημένη μας πρόταση και στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους μεταξύ αυτών και εσάς. Ο στόχος είναι να υποβάλουμε καινούρια πρόταση πριν το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου έτους. Και βέβαια εσείς θα συμμετάσχετε στενά. Περιμένω να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Αυτά, Πρόεδρε, θα κάνω μια παύση. Έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά θα πρέπει να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Βεβαίω σας ευχαριστούμε εμείς Επίτροπε Μάλστρομ για την παρουσίαση του πρόγραμματος εργασιών, για την ενημέρωση όσον αφορά την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών 2011 και για την συνεχή ετοιμότητά σας να συνεργάζεστε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εμφανιζόμενοι εδώ και ανταλλάσσουσα απόψεις μαζί μας όσο συχνά χρειάζεται και όποτε είναι δυνατόν. Έχουμε 21 μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο και έχουμε μία ώρα μπροστά μας, στη διάθεσή μας, μία ώρα, οπότε προτείνω να γίνει ένας πρώτος γύρος συντονιστών, τρία λεπτά, και μετά τα υπόλοιπα μέλη θα υποβάλουν τις ερωτήσεις τους ή θα κάνουν τα σχόλιά τους, ένα δίλεπτο καθένας, διότι και ούτω τρόπο θα έχουμε και κάποιο χρόνο να μπορεί να δευτερολογήσει η Επίτροπος, να απαντήσει μάλλον η Επίτροπος. Κλείνουμε τον κατάλογο, 21 μέλη έχουμε. Πρώτο γύρο για του συντονιστέ και ξεκινά ο κύριο Μπουσετήρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ εκ νέου και που ήρθατε εδώ με καλές ειδήσει όσον αφορά τις άκρο ενεργητικές ε, πρωτοβουλίες που αναλάβατε. Το εκτιμούμε τα μάλα στην Επιτροπή μας, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε απαραίτητα όλων, αλλά σίγουρα έχετε την υποστήριξή μας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που προτείνατε, κυρίως όσον αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση που ε, υποβάλλατε πρόσφατα. Είναι μια πολύ καλή και ισορροπημένη πρωτοβουλία αυτή. Προσβλέπουμε να διαβάσουμε αναλυτικά αυτά που ξεκινήσατε σήμερα. Δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό, απλώς αναφέρατε κάποια σημεία. Προσβλέπουμε λοιπόν ε, στην ανάλυση των λεπτομεριών αργότερα. Το Σέγγεν, σας υποστηρίζουμε όταν λέτε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε το σύστημα του Σέγγεν και θέλω αυτό εκ νέου να το ξεκαθαρίσω, το είπαμε στη συζήτηση, το λέμε ξανά σήμερα. Όμως, νομίζω ότι αυτό που μάθαμε από τις πρόσφατες δυσκολίες όσον αφορά τα σύνορα Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελεύθερη Ευρώπη άνευ σύνορων θα πρέπει να δεχθούμε ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι κοινή μερίμνα, κοινή φροντίδα. Διότι τελικά τα εξωτερικά σύνορα είναι η πηγή των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας ή σε άλλες περιπτώσεις επίσης. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση, δηλαδή μεταξύ Ευρώπη που δεν έχει εξωτερικά σύνορα από τη μια και εξασφάλιση των εξωτερικών σύνορων από την άλλη και συλλογικά να επομιστούμε την ευθύνη κάνοντα το αυτό. Οπότε έρχομαι τώρα στο θέμα τη αλληλεγγύη. Πριν έρθετε, κύριε Επίτροπε, είχαμε μια παρουσίαση μια εκθέσεω, μια μελέτη όσον αφορά το άρθρο 80 των συνθηκών περί αλληλεγγύη και δίκαιου, δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών. Θα θέλαμε να τη δείτε και να εφαρμόσετε αυτό το άρθρο γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο για μας. Πρόσφατα κατόπιν δικής της προσωπικής πρωτοβουλίας παροτρύνατε όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την αλληλεγγύη συγκεκριμένα. Αλληλεγγύη με χώρες όπως η δική μου και ετοιμάσατε με διάσκεψη παροτρύνοντας ε, τα κράτη-μέλη να δεχθούν τον ε, παναπατρισμό, ανέλαβαν, μετακίνηση μάλλον, κράτη-μέλη δέχτηκαν να πάρουν 323 ε, μετανάστες και να πάρουν τους μετανάστες από τη Μάλτα και να πάνε σε άλλα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία. Την επόμενη μέρα, όπως το ήξερα, ένα σκάφος με 350 άτομα ε, διεσώθη στην ανοιχτή θάλασσα. Και όλη αυτή η δουλειά που κάνατε, πριν αυτή την πρωτοβουλία ε, για την αλληλεγγύη, καταστάθηκε την επόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται ένας μόνιμος μηχανισμός με ένα βαθμό αυτόματης λειτουργίας που να μπορεί να ξεκινά και να μην χρειάζεται επίτροπος να απευθύνει εκκλήσεις στα κράτη-μέλη κάθε φορά. Και εδώ χρειαζόμαστε την ε, αλληλεγγύη. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι προσβλέπουμε στις πρωτοβουλίες σας για τα θέματα που θίξατε, όπως το σύστημα εισόδου-εξόδου το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Χρηματοδότηση των, Τρομοκρατών. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που είπατε και επίσης ε, μας ενδιαφέρει και η πρωτοβουλία σας για τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ε, είπαμε τρία λεπτά. Ο κύριο Μωράης, εσεί συμμορφωθήκατε, είστε πολύ καλό. Είστε παράδειγμα ο κύριο Θα προσπαθήσω να μιλήσω λιγότερο από τρία λεπτά, λέει ο κύριο 20 συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν, οπότε θα είμαι πραγματικά σύντομο. Και έχω το μάτι στραμμένο στο ρολόι. Μπορούσα λοιπόν να πω καταρχά, ε, κύριε Επίτροπε, σας χειροκροτήσαμε γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε τεράστιο όγκο ανακοινώσεων πολιτική ε, πίεσης, ε, όλα αυτά. Τώρα για να επιστρέψω στην ουσία της υπόθεσης για την ομάδα μας. Εάν βγάλουμε όλα τα πολιτικά ζητήματα. Το Σέγγεν είναι ουσιαστικά ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υπάρχουν ε, εξωτερικά σύνορα. Ξεκινάμε τώρα το θέμα της ε, λαθρομετανάστευσης, των σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Ακόμα δεν υπάρχει δηλαδή ε, πολιτική, πολλά ακόμα είναι τα εκκρεμή νομοθετικά ζητήματα. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω στους αδέλφους και τους Σάιμον κυρίως, ότι εάν πρόκειται να υπάρξει ένας ε, κοινό μηχανισμός burden sharing με ελληνική, καλό θα ήταν να σταματήσουν ε, οι αντιδράσεις και κυρίως επίπεδο συμβουλίου και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καιρό πιστεύετε ακόμα ότι θα αντιστέκεται στο θέμα αυτό το συμβούλιο, πόσο θα, μπορεί, θα προσπαθεί ακόμη την νόμιμη μετανάστευση να την κατακαιρματίσει σε ε, θεματικέ ομάδε. και φυσικά πρέπει να επισημάνω εδώ ότι δεν έχω καμιά αμφιβολία πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λύσει ουσιαστικά τα αισθήματα αυτά και θα ήθελα να σα χαρώ επί τη ευκαιρία για τι προτάσει σα σχετική με την πολιτική γειτονία σα. μόλι άρχισα την ανάγνωση των προτάσεων αυτών τεράστιο έργο και θα συγχαίρω. Θα ήθελα όμω να επανέλθω με το κύριο ζήτημα που έχουμε ω ομάδα. Ξεκινήσατε με φιλόδοξες ε, προτάσεις, η παραδείγματι προτείνεται εταιρική σχέση με χώρε που έχουν κάποιες ε, οδούς, κάποιες λύσεις νόμις μετανάστευσης, η συνεργασία αυτή να ε, ενισχυθεί. Το Συμβούλιο όμως αντιστέκεται. Δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε ε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, γιατί δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πουθενά. Μέχρι το 2012 δεν θα έχουμε λύση αν δεν κινηθεί και δεν αλλάξει θέση στο Συμβούλιο. Ξέρουμε το θέμα αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει πολύ, δεν πρόκειται να προχωρήσει ως έκθεση πρωτοβουλίας από το Κοινοβούλιο, αλλά αν πρόκειται να υπάρξει νομοθετική πρόταση, παρακαλώ ενημερώστε μας για να ετοιμαζόμαστε και εμείς για να γνωρίζουμε και τι είδους ε, θέσεις μπορεί να εκφράσει το Κοινοβούλιο ή τι είδους μάλλον ε, συμμετοχή στη δικασία αυτή μπορεί να έχει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντο. Η κυρία Γκόμπερ, το κοινοβουλιο ευχαριστω πολυ Κλόντα. ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Έχετε επισκεφτεί την Επιτροπή μας ως 10 φορές και περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω για την παρουσία σας εδώ. Κάθε φορά με ιδιαίτερη απόλαυση ε, συνεργαζόμαστε μαζί σας ε, και ακούμε τις παρατηρήσεις σας, τις απαντήσεις σας. Ελπίζουμε και οι λοιποί επίτροποι να επιδείξουν έστω και το ίμιση της δικής σας δραστηριότητας και αποφασιστικότητας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί ως προς τα όσα διαπιστώνουμε και τόσο διεκδικούμε. Διαπιστώνουμε οικονομική κρίση, ακόμη στην Ευρώπη ε, κρίση η οποία οδηγεί σε, σε λαϊκιστικές αλλά ακόμη και άκρες λαϊκιστικές εξάρσεις. Ακόμη και τώρα υπάρχουν προσεγγίσεις από ορισμένε κυβερνήσεις πτυχών που δεν αναμέναμε να αντιμετωπιστούν κατά αυτόν τον τρόπο πριν από 4-5 χρόνια με πρόσχημα, σαφρό μάλλον, γελίο θα έλεγα. Δεν αντιμετωπίζουμε μαζικέ μεταναστευτικέ ροέ, επειδή ήρθαν κάποιοι, ε, επειδή ξεσηκώθηκαν κάποιοι στη Βόρεια Αφρική να διεκδικήσουν την ελευθερία του. Απλώ κάποιοι αναζητούν από τράγους τράγου και δυστυχώ οι λύσει που δόθηκαν σε ορισμένε περιπτώσει ήταν κάκιστε. Ταυτόχρονα σας βεβαιώ ότι έχετε την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής μας και γενικότερα του Κοινοβουλίου πιστεύω όταν ε, τίθεται ζήτημα των ε, προτάσεων μέτρων για το άσυλο και την ε, μετανάστευση και θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πρόθεσή μα να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε ένα πακέτο συνολικό, σε, ένα, σε μια κάλυψη ε, των νομοθετικών ε, ζητημάτων στο σύνολό του, γιατί για μένα είναι πολύ δύσκολο διαφορετικά να ε, δεχθώ την Ευρωπαϊκή Ένωση ω παράγοντα διεθνή, εάν δεν δράσουμε όλοι μαζί και οι 27. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και αισιόδοξη ως προς, το, προς την δεκτικότητα του Συμβουλίου στο θέματα αυτά. Τούτου λεχθέντος, δεν θέλω να φερθώ στο ζήτημα του Σέγγεν και σε ζητήματα που έχουν, επί, ε, έχουν ε, εγερθεί και στο παρελθόν. Στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα και με ισχύουσα τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να επανεισαγάγουν για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα τον, τους ε, μεθοριακούς ελέγχους και γνωρίζω βεβαίως ότι δεν βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την ίστατη στιγμή που σημαίνει ότι ε, έχουν παραλυφθεί κάθε μορφή έλεγχη από πλευρά Επιτροπή ε, και Κοινοβουλίου και ότι παραγνωρίζεται πλήρω η κατάσταση. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξή. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση ή απλώ ανοίγουμε την ε, θύρα σε νέου μηχανισμού που θα οδηγήσουν σε μια ίστατη λύση αυτού του τύπου. Γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώ προ τα πού κινούμαστε. Επίση, θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και είχα την εντύπωση ότι η διαφθορά θα έπρεπε μάλλον να υπάγεται στην, ε, στον τομέα της δικαιοσύνη. Βλέπω όμω ότι εσεί έχετε επιληφθεί της καταπολέμησης της διαφθοράς. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Για το UTFTP δεν, ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είδου επιλογές θα προκύψουν. Η τρίτη επιλογή με ανησυχεί μάλλον, γιατί αν είναι μεικτό το σύστημα νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορεί να χαθούν ε, και να βρεθούν εκτός ελέγχου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Φλότφα. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη διάθεσή της να έρθει εδώ να μας μιλήσει για τις διάφορες πρωτοβουλίες ε, που μπόρεσε να αναλάβει σε ένα τόσο διαφιλονικούμενο ε, και συγκρουσιακό θέμα στο οποίο εκφράζονται πολλές φορές οι εθνικοί εγωισμοί και η εθνική μοιοπία έναντι του ευρωπαϊκού οράματο. Θα ήθελα λοιπόν, χωρί να έχω τη δυνατότητα ακόμη, χωρί να έχω αποκτήσει ακόμη τη δυνατότητα να εξετάσω αυτέ τι προτάσει, ε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ανακοίνωση σχετική με την εισαγωγή μέτρων για τι επιπτώσει ε, των εξελίξεων στη νότια όχθη τη Μεσογείου, γιατί πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση στη σχέση μα με αυτέ τι χώρε, Στο συνότιο όχθη τη Μεσογείου μπορεί να ε, αποτελέσει μια ευκαιρία και για ανταλλαγέ και για κινητικότητα, ταυτόχρονα βλέπω ότι ε, χειρίζεστε το θέμα αυτό με τα κλασικά μέσα της πολιτικής μας, δηλαδή αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λαθρομετανάστευσης. Επομένως, η τυποποιημένη αντίδραση μέσα από το έγγραφο είναι πολύ επιθυμητή βεβαίως και ευκταία, πλην όμω διαπιστώνω ότι δυστυχώ το οπλοστάσιο το οποίο τη συνοδεύει μάλλον θα μα απαγοητεύσει γιατί ε, έχουμε ήδη στην περιοχή αυτή την εφαρμογή μέσων και νομοθετημάτων που ήδη ισχύουν, είναι πολύ γνωστά. Δεν βλέπω καμιά διαφοροποίηση, φυσικά αυτό ελέγχεται, αλλά δεν βλέπω καμιά καινοτομία ως προς τη δική σας προσέγγιση, μια καινοτόμο προσέγγιση στα, σε σχέση με την περιοχή αυτή. Αλλά ίσως και να υποτιμώ ε, την, τις, τους χειρισμούς σας και τις επιλογές σας. Πρέπει να τα μελετήσω πιο προσεκτικά. Και βέβαια θα ακούσω και τις απαντήσεις σας με μεγάλη προσοχή. Επίσης, ζητήματα τα οποία έχουν εδρεωθεί, πιστεύω, και αποδειχθεί με πολλά αποδεικτικά στοιχεία, ε, το πόσα δηλαδή μπορεί να συμβάλλει στα, στο κοινωνικό κόστος στα κράτη-μέλη ή μετανάστευση, είναι ζητήματα τα οποία ε, θα πρέπει να συζητήσουμε εν ώψη μιας τοποθέτησης γενικής και πολιτικής επιλογής εναντί της μετανάστευσης. Εγώ έχοντας την ευκαιρία να συζητήσω ε, τα θέματα αυτά στη Γαλλία σε μια συζήτηση τρογγυλής τραπέζι με παρουσία πολλών και γερουσιαστών Γάλλων συναδέλφων ε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι συνολικά οι μετανάστες προσφέρουν στο κοινωνικό ε, σύστημα των κρατών της Γαλλίας συγκεκριμένα 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτό με ό,τι άλλο κόστος μπορεί να υπάρχει και όταν έχουμε να κάνουμε με τις μεγάλες ανισότητες και τις ανισορροπίες του κοινωνικού κόστος θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για την ε, επιχείρηση Rabbit στην Ελλάδα. Ε, πήγα να συστήσω με τους ανθρώπους της επιχείρησης αυτής και μου είπαν ότι δεν αλλάζει τελικά ο αριθμός των αφικνουμένων στην Ελλάδα. Μπορεί στο συγκεκριμένο αυτό κομμάτι ε, των συνόρων να περιορίζονται οι ροές, αλλά στα 20 χιλιόμετρα πιο κάτω ε, αλλάζουν προς τα πάνω οι ροές, Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν να περάσουν από πάνω τώρα περνάνε από πιο νότια. Και ω εκ τούτου δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα δηλαδή από το σύστημα. Και γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε και λίγο πιο ορθολογιστέ, λίγο πιο πρακτικοί και λίγο πιο λογικοί ω προ την ε, εισαγωγή ε, προδεδικασμένων ε, ιδεών ε, και ιδεοληψιών περισσότερο για το θέμα της μετανάστευσης. Και θέλω να ρωτήσω αν σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλία ως προς τους μόνους και ανήλικους μετανάστες, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δραματική, αλλά και παρουσιάζονται πολύ διαφορετικές εικόνες της κατάστασης που γνωρίζουν οι νέοι ανήλικοι που ζουν μόνοι τους στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Σταβάρης. Ο κύριος Σταβάρης. Ευχαριστούμε που μας επισκέπτεστε δεύτερη φορά σήμερα. Θα ξεκινήσω με τη Σέγγεν. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στη στάση μας έναντι οποιασδήποτε πλαστής πίεσης ε, επί της Σέγγεν. Γιατί οι πιέσει αυτές είναι πιέσει εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να βλέπει να πλήττονται και οι δύο σημαντικοί πυλώνες της, το ευρώ και η Σέγγεν, ταυτόχρονα. Και να βρίσκεται σε οικονομική κρίση, ταυτόχρονα. Συνεπώς, οι οπορτουνιστικές, επιλεκτικές, μονομερείς αποφάσεις για κλείσιμο συνόρων και για επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι ε, να καταλήξουν να είναι συστημικές. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στις κυβερνήσεις ε, να ασκούν κοινική πίεση επί της Συμφωνίας Σέγγεν. Γιατί η συγκυρία θα μπορούσε να είναι πολύ θετική για θέματα όπως οι μεταναστευτικές ροές, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Είμαστε στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου κόσμου. Είμαστε στη μετάβαση. Από ένα κόσμο στον οποίο ε, είχαμε αναθέσει τη βρώμικη δουλειά που θέλαμε εμείς να κάνουμε στον Καντάφη και στους διάφορους Καντάφιδες, τελειώνει αυτός ο κόσμος. θα πρέπει να ακολουθεί ρεαλιστική προσέγγιση στην μετανάστευση και στη σχέση μας με τις γειτονικέ χώρες. Χτες ε, συναντήθηκα με έναν σημαντικό Πορτογάλιο ιστορικό που μου έλεγε ότι στο ερευνητικό του κέντρο δεν μπορεί να έχει ερευνητέ από το Μαρακές, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να καλέσει ούτε ένα πρίτανη από την άλλη μεριά της, από την άλλη όχθη της Μεσογείου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η προσέγγιση μας θα είναι ορθολογική, αλλά και ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε την άλλη όχθη της Μεσογείου με περισσότερες πολιτιστικές και προσωπικές ανταλλαγές. Μετά, για το πακέτο ασύλου. Χρειάζονται πιο γενναίες προτάσεις από πλευράς Κομισιόν. Η στρατηγική ήταν η σαλαμοποίηση του πακέτου με προώθηση των πιο εύκολων κομματιών. Ενώ τα πιο γενναιόδαρα τμήματα τα αφήναμε για αργότερα. Όμως αυτό αμφισβητεί το ίδιο το πακέτο το ολόκληρο. Μετά, η επανεγκατάσταση. Ε, νομίζω ότι δεδομένου ότι έχουμε το πακέτο, το, πιλο, το πιλωτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά. Θα ήθελα να μου πείτε ε, ποια διδάγματα έχετε εσείς πάρει από την παρακολούθηση της εφαρμογής του, ε, πακέτου, του προγράμματος SWIFT για την ε, πήγουσα επανεγκατάσταση. Πρόεδρος, ε, παρόλο ότι είχαμε κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών, βλέπω καινούργια χέρια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ελαστικοί γίνεται, όσο πιο ανοιχτοί γίνεται, αλλά έχουμε και κάποια χρονικά όρια. Όρο λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Αλλά, όρος είναι να ε, τηρούμε τους χρονικούς περιορισμούς. Κύριος Κλέης. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ανησυχώ. Και ανησυχώ διότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής δημιουργούμε την εντύπωση ότι δημιουργούμε πλαστά οικοδομήματα. Από συναντήσεις με κάποιους συναδέλφους φαίνεται ότι υπομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα. Και υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της επίσημης Ευρώπης από τη μια και τους πολίτες από την άλλη. Υπάρχει αυτό το, η διαφορά μεταξύ του δρόμου και Στρασβούργο. Το ότι γίνονται έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, το ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι ε, βλέπουμε το θέμα από την άλλη πλευρά ότι μιλάμε για την εισαγωγή νέων εσωτερικών ελέγχων και αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Όχι, ο λόγος είναι διαφορετικός. Το πρόβλημα είναι ότι το Σέγγεν δεν λειτουργεί. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μεν, αλλά δεν διενεργούνται ενεργούνται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα δε. Εκεί έγκυται το πρόβλημα και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπόρεσα να δω ότι είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σημαντικά θεμελιώδη βήματα που απαιτούνται. Ακούμε αναφορά σε τάσεις ε, στα κοινοβούλια, ε, διάφορες λαϊκιστικές δυνάμεις που ανέρχονται σε δύναμη, αλλά κοιτάξτε ποια είναι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ποιε επιλογέ υπάρχουν στο Σέγγεν. Μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσει μπορούν να επανέλθουν εσωτερικοί έλεγχοι. Αν υπάρχει τρομοκρατική απειλή, αν υπάρχουν αθλητικέ εκδηλώσει, αν απαιτείται αυτό, να υπάρχουν εσωτερικοί έλεγχοι, διότι ίσω δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Αν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για εσωτερική μετανάστευση, τότε ε, θα πρέπει να επαναφερθούν αυτοί οι έλεγχοι και να διενεργούνται γρήγορα. Από ό,τι μας είπατε κύριε Επίτροπε, εγώ δεν κατάλαβα ότι είσαστε έτοιμοι να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, ερώτημα. Πρακτικά, τι βήματα θα προτείνετε εσείς. Πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορούν τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με έγκαιρη προειδοποίηση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουν τα σύνορά του, ακόμα και αν δεν είναι αυτά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θέλετε να απαντήσετε στου συντονιστέ πριν προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία. Ναι, ίσω ε, θα μπορούσα να το κάνω. Και ίσω εξαφανιστούν κάποιε ερωτήσει αν απαντήσω σε αυτά που υπόθηκαν τώρα. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ και για τη σημότητα όλων των ομάδων να ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν μετανάστευση και τα σύνορα και να ακολουθεί μια συνεχτική προσέγγιση, διότι όπω πολύ είπατε, είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να πέσει κανεί στην παγίδα ότι υπάρχουν υπεραπλουστευμένε λύσει. Δεν υπάρχουν τέτοιε. Είναι όλα πάρα πολύ περίπλοκα και όλα πάνε μαζί. Πρέπει να το δούμε μακροπρόθεσμα. Χρειάζεται να ηγηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπέσουμε στην παγίδα σύμφωνα με την οποία η λύση είναι να κλείσουμε τα σύνορα και όλα είναι μια χαρά ε, περνάμε δύσκολους καιρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να το πω αυτό. Και θα έχουμε τεράστιε δυσκολίε όσον αφορά πολλά από αυτά τα θέματα. Όσον αφορά του ελέγχου στα σύνορα, κύριε Μπουσετήλ, βέβαια τα κράτη-μέλη υπέχουν υποχρέωση ελέγχου των σύνορων. Αυτό είναι και το νόημα του κράτου. Εφόσον υπάρχουν και κοινά σύνορα, υπάρχει και πολύ μεγάλη ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Και ελπίζουμε ότι ο κανονισμό για το Frontex θα εφαρμοστεί σύντομα, θα είναι έτοιμος γιατί το ετοιμάζουμε μελέτη βιωσιμότητας για κάποιο μηχανισμό ευρωπαϊκό ελέγχου των συνόρων και γι' αυτό ελέγχουμε και το μηχανισμό αλληλεγγύης. Με τα χαράς να δω το έγγραφο που σας παρουσιάστηκε πριν καταφτάσω εγώ. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δείξουν αλληλεγγύη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδε. Μπορούμε να βρούμε διάφορα κίνητρα να δώσουμε διάφορα μέσα. Αλλά δεν μπορείτε να υποχρέσετε τα κράτη-μέλη να είναι αλληλέγγυα. Και κάποια κράτη-μέλη ε, δεν δέχτηκαν ε, κανένα πρόσφυγα ούτε από τη ΜΑΤΑ ούτε από το κατάλογο της ΥΠΑ της Αρμοστίας πρόσφυγης του ΟΗΕ. Εάν υπάρχει σύστημα ασύλου τότε θα υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να μοιράζονται την ευθύνη για τους ετούντε άσυλο που έχουν. Διότι 10 χώρες σήμερα παίρνουν το 90% των ετούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχουν άλλες χώρες που θα μπορούσαν πιθανότατα να κάνουν κάτι περισσότερο. Ο κύριος Μωράης, συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά το πακέτο για το άσυλο. Γι' αυτό προσπαθούσαμε τόσο πολύ ε, να μείνουμε μαζί, να μην κάνουμε το γύρο DAC, εάν δεν υπάρξει πρόοδο σε άλλους τομείς αυτή είναι η θέση που περασπίζομαι έναντι 27 κρατών μελών ε, στο Συμβούλιο. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης του μηνός ε, θα δώσει όθηση στο θέμα. Θα έχουμε έναν οδικό χάρτη που θα ετοιμαστεί και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη, οι αρχηγοί κατών κυβερνήσεων να εγκρίνουν τον οδικό χάρτη και να πιέσουν τους υπουργούς εσωτερικών να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Διότι όλα τα κράτη-μέλη, με ελάχιστε εξαιρέσεις, ε, λένε ότι δεν θα είναι έτοιμα ε, πριν το 2012. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά είναι η μόνη προσέγγιση. Για την ε, ολοκλήρωση δεν υπάρχει νομοθετική πρόταση, υπάρχει ανακοίνωση που αναφέρεται στις βέλτιστες πρακτικές, δείκτες, μοντέλα, συλλογή στατιστικών κλπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υπάρχει συνεισφορά, αλλά οι Βρυξέλλε δεν μπορούν να εντάξουν του μετανάστε. Αλλά μπορούμε να το θέσουμε σαν ένα θέμα στο, στην ευρωπαϊκή ατζέντα, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το Σέγγεν. Πρέπει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Πρέπει να βελτιώσουμε την αξιολόγηση και τον έλεγχο και του μηχανισμού και αυτό θα πρέπει να γίνει επικοινωτική βάσεω πρέπει να φεύγουμε, όχι να φεύγουμε, να αποτιμήσουμε όλα τα εργαλεία που ε, μπορούν να διατεθούν στα κράτη-μέλη όταν έχουν ένα πρόβλημα και πολύ έγκαιρα. Ε, θα πρέπει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε συστάσει και κατευθυντήριε γραμμέ σχετικά με το πώ θα ερμηνεύονται τα διάφορα μέτρα. σω ενδεχομένω υπάρξει ανάγκη διευκρίνηση. Πότε σε εξαιρετικέ περιστάσει τα κράτη-μέλη μπορούν να δράσουν πέρα από αυτά που προβλέπονται ήδη Είδαμε τις περασμένες εβδομάδες υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που ερμηνεύουν το κεκτημένο Σέγγεν πολύ ευρύτερα από ό,τι ήταν η πρόθεση των συντακτών του κειμένου. Αν αλλάξει κάτι εκεί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθηθεί κοινοτική προσέγγιση, να είναι κοινή α, απόφαση, να μην κάνει κάποιο κράτος στα δικά του. Πρέπει να δούμε υπάρχει ρεαλιστική προσέγγιση, θα το πετύχουμε αυτό χωρίς να ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου και αποδυνάμωση του Σέγγεν. Μπορούμε να ενισχύσουμε το μηχανισμό που ήδη υπάρχει για τη διακυβέρνηση και την εποπτεία και ίσως να το πετύχουμε αυτό. Κινητικότητα. Σύμπραξη, συνεργασία πάνω σε αυτό, κυρία Φλότρο. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι κάπως καινούριο, προσπαθώντας όλα αυτά τα στοιχεία να τα έχουμε στη διάθεσή μας και να συζητούμε ανοιχτά καινοτόμα με τα νέα καθεστώτα αυτών των χωρών. Ελπίζουμε νέα καθεστώτα, υπάρχουν κάποια προβλήματα, ξέρετε, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργασία ευρεία, συζητώντας ανοιχτά, χωρίς προκαταλήψεις. Θα τα καταφέρουμε, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά είναι η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιδοθεί σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό κρύβεται πίσω από την ανακοίνωση που υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τους απομονωμένους ανηλίκους δεν υπάρχουν νέες ε, δρομολογηθείς πρωτοβουλίες αλλά κάνει μια αποτίμηση κάθε χρόνο το Συμβούλιο και στις προτάσεις του πακέτου ασύλου αναφέρεται ειδική προστασία για τους απομονωμένους ανηλίκους και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μην εξαφανιστεί αυτή η αναφορά και στην οδηγία για το εμπόριο ανθρώπων υπάρχουν διατάξεις που δεχθήκατε που προστατεύουν ειδικά αυτές οι κατηγορίες των ευάλωτων παιδιών. Πρόεδρε, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Ότι κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος, ξεκινάμε ένα δεύτερο γύρο. Να σας πω, κυρία Επίτροπε, διότι αναφερθήκατε, σχολιάσατε την παρουσίαση που, κάνα, που είχαμε από τον καθηγητή Βαν Χόιλε για τη ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 80 και το τι υπετίθετο, τι, τι εστήριζε αυτή την παρουσίαση. Κάτι που ζήτησε η Επιτροπή μας. Ότι δεν θα υπάρχει ρήτρα αλληλεγγύης μέχρι να κατανοήσουμε πλήρως ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνα θα υπάρχει κάτι δεσμευτικό. Δεν θα υπάρχει ρήτρα για αλληλεγγύη αν δεν υπάρχουν θεσμικές ρυθμίσεις και περιεχόμενο. Ότι θα είναι δεσμευτικός νόμος αυτός περί αλληλεγγύης. Πολλά συντάγματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι συντάγματα τα οποία ε, εφαρμόζονται σε αποκεντρω... με ε, σε αποκεντρωμένες χώρες που προβλέπουν στην εσωτερική ένωμη τάξη αλληλεγγύη. Αλλά αυτή η αλληλεγγύη δεν θα έχει οδήποτε πρακτικό νόημα αν δεν υπήρχε θεσμική διευθέτηση που θα εξυπηρετεί την εφαρμογή αυτού του μέτρου δεσμευτικά. Τι σημαίνει στην πράξη ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την ερμηνεία της αλληλεγγύης στην ελεύθερη βούληση των κρατών μελών, διότι αυτό δεν θα ήταν αλληλεγγύη, θα ήταν ελεημοσύνη, αδερφοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκύτητα ε, όσον αφορά τη γεωγραφική γειτονιά κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, δεν θα ήταν όμως πραγματική αλληλεγγύη. Συνταγματικά θα πρέπει νομικά να καλύπτεται και να ορίζεται. Μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος, αλλά αυτό είναι ένας οδικός χάρτης. Ε, θα πάρει χρόνο, αλλά είναι ένας οδικός χάρτης. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε επόμενους ομιλητές. Σας παρακαλώ όμως να περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο ούτως ώστε να υπάρξει δεύτερο γύρος απαντήσεων της Επιτρόπου Μάλστρομ, ξεκινώντας από τον κύριο Δίας Δεμέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν προς την Επίτροπο. Το έργο της είναι απαραίτητο πολύ καλά καμωμένο και η ανακοίνωσή της πραγματικά πολύ βάσιμη. Αναγνωρίζονται καταρχήν οι μαζικές ε, μετακινήσεις πληθυσμών, 650.000 ατόμων. Ευχαριστώ πολύ για την ορολογία που χρησιμοποιείτε, που είναι η πιο κατάλληλη. Ε, αυτή που είναι παράνομη είναι η, ε, τα κυκλώματα. Τα άτομα δεν είναι παράνομοι μετανάστες, είναι λάθρο μετανάστες. Ε, αυτό το έχει πει το Κοινοβούλιο επανειλημμένο στο παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ που αναγνωρίζετε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, ούτε επαρκώς εξοπλισμένη για να αντιμετωπίζει κρίσει τέτοιου μεγέθους όπως αυτή της Βόρειας Αφρικής. Ευχαριστώ επίσης που αναγνωρίζετε ότι τα τέσσερα ταμεία είναι ανεπαρκή και επιπλέον δεν μπορούν να κινητοποιηθούν εύκολα. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε και να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη και στην πράξη αλλά και νομικά. Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε πως ε, το μεγαλύτερο τμήμα των λαθρομεταναστών ε, είναι άτομα τα οποία έχουν ξεπεράσει το χρόνο νόμις διαμονής που προβλέπεται από την θεώρησή τους. Ευχαριστούμε επίσης που είστε υπέρ της διεθνούς προστασίας ε, και της ένταξης των μεταναστών. Ε, το, η ανακοίνωση σας έχει δύο σημαντικά ε, στοιχεία. Πρώτον, οι πρωτοβουλίες οι οποίες συνδέονται με την ε, ανακοίνωση που είναι 32 και εκ των οποίων τέσσερις ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ευχαριστούμε πολύ και για τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δίνετε, πολύ σημαντικά. Για τη Σέγγεν, με δύο λόγια. Κατά την άποψή μου η Σέγγεν πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να υπεραμεινθούμε τη Σέγγεν και θα πρέπει η Σέγγεν να είναι, και μάλλον και πρέπει πάντοτε η λύση οποιαδήποτε κρίση να είναι κοινή, όχι μοναχική. Και τελειώνω λέγοντας ότι ο κ. Μπουσουτήλ μόλις μου είπε ευτυχώς πως το Κοινοβούλιο ε, έλαβε ε, άδεια να στείλει μια αποστολή στα σύνορα μεταξύ Λιβύας και Τινησίας για να κάνει εξολόγηση κατάστασης. Ευχαριστώ δεν σας ζηλεύω, Επιτροπή, με όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρή κατάσταση την αμφισβήτηση του κεκτημένου του Σέγγεν, της απελευθέρωση από την υποχρέωση για θεώρηση διαβατηρίων, περαιτέρω επέκταση του Σέγγεν. Είπατε κι εσείς σήμερα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών χάρη στο Σέγγεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα έλεγα ότι για τα Δυτικά Βαλκάνια ιδιαίτερη σημασία είχε το καθεστώς, η απελευθέρωση μόνο το καθεστώ υποχρέωση ε, θεώρηση. Τώρα, ε, μιλήσατε νωρίτερα για την δυνατότητα, η πιθανότητα προσωρινή άρση αυτή τη ε, απελευθέρωση. Με χαρά σημειώνω την παρατήρηση ότι αυτό θα συμβεί σε άκρος εξαιρετικέ περιστάσει μόνο. Το σημειώνω λοιπόν. Αλλά θα ήθελα να πω και το εξή ότι διαβάζω στο κείμενο, δεν είμαι βεβαία εάν πρόκειται για μια αυτόματη απόφαση ή εάν θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό ε, μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής Κοινοβουλίου και μετά να ληφθεί μια απόφαση για την άρση της υποχρέωσης. Επίσης, έχουμε ιδιαίτερα για την Σερβία και τη Μακεδονία, πολλούς ψευτοετούντες άσυλο. Ε, έχετε κάποιες ε, πληροφορίες τελευταίες, γιατί είχαμε ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε μια κινητικότητα των κυβερνήσεων των κρατών αυτών ε, προκειμένου να λάβουν μέτρα και να αντιμετωπίσουν αυτέ τι ψεύτικε αιτήσει, τι ε, ψευδεί αιτήσει. Μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα με, με σοβαρότητα την ενάρξη των διαπραγματεύσεων για την άρση της υποχρέωση θεώρησης με το ψηφοπαίδιο όπου ξέρω από τις συνομιλίες που είχα μαζί τους ότι αισθάνονται μεγάλη δυσφορία διότι δεν ξέρουν πώς να χειριστούν το θέμα από πλευρά τους. Καλό λοιπόν θα ήταν ε, οι κυβερνήσεις να γνωρίζουν ακριβώ τι θα πρέπει να κάνουν και είναι απο μονομένο το κοσφοπέδιο που τελικά υποχρεούνται οι πολίτες του να αναστήσουν λαθρέους τρόπου να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πλαστά-πλαστό ε, διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και εκεί πέρα νομίζω θα πρέπει να ε, δούμε την πραγματική ουσία του προβλήματος. Κυρία Λάτφορντ, Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαια ότι ένα τόσο, μια τόσο μεγάλη πρόκληση, ένα τόσο δύσκολο ζήτημα, μόνο στα δικά σας ικανά χέρια θα μπορούσε να βρει λύση. Πάντω η κατάσταση είναι κάπω δύσκολη, αυτό που το ομολογούμε πιστεύω και όταν ε, πριν από κανένα δύο εβδομάδε συζητήσαμε πάλι, είχατε υπογραμμίσει τη στράτευσή σα, στράτευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προστασία του χώρου του Σέγγεν και τη ελεύθερη κυκλοφορία χωρί σύνορα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα σε αντιπαράθεση όμως με την πληθώρα σχολείων που μεταφέρει ο τύπος ε, τα οποία σχόλια δίνουν την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βρει μία απλουστευμένη ευχερέστερη μορφή επανεισαγωγής των ελέγχων στα σύνορα. Εξού θα έπρεπε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα γιατί νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό σημαίνει ουσιαστικά κοινοτικοποίηση τη διακυβερνητική μεθόδου, του διακυβερνητικού μηχανισμού. Θα ήθελα να σα επισημάνω τον κίνδυνο τη λεξούλα εισάγει. Γιατί ήταν η λέξη εισάγει, αυτή η μικρή λέξη στη σελίδα 8 τη ανακοίνωσή σα και στη σημερινή, στο σημερινό κείμενο, της εισαγωγής μιας ασφαλιστικής ρήτρα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άλλες ερμηνείες. Βέβαια εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν ε, οι κρίσιμες περιστάσεις, οι εξαιρετικές περιστάσεις, οι σπάνιες περιστάσεις, το το προσδιορίσατε αυτό και είπατε ρητά ότι ε, πιστεύετε ή ελπίζετε ότι χρειαστεί ποτέ να εφαρμοστεί αυτή η διασφαλιστική θα δικλίδα που θα επαναφέρει την υποχρέωση για του διαβατηρίου. Αλλά ο τύπο διαβάζει διαφορετικά αυτή τη λέξη. Το εισάγει και ω εκ τούτου, εάν μου επιτρέπετε να διατυπώσω μια πρόταση, μια συμβουλή, θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές, στο βαθμό που μπορείτε βέβαια, ε, το κείμενο έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν να παρερμηνεύσουν οι δημοσιογράφοι, αν και έχουν την τάση εν γέννη, τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ουσία της υπόθεσης αυτής, δηλαδή την ε, περίπτωση ή μη επανεισαγωγής ελέγχων στα σύνορα και θεώρησης διαβατηρίων. Η μη Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ και θεωρησης διαβατηριων κυρια κελλερ επίσης ε, διότι βλέπω ότι το Σέγγεν ε, μαζί με την απελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίων είναι θέματα επίκαιρα για σας και πρέπει να παραμείνουν όπως είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό συμφωνούμε και για την κυρία Φάζο νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα στο θέμα της απελευθέρωσης από το καθεστώς ε, της θεώρησης διαβατηρίων πώς θα μπορέσουμε εμείς δε, ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ των πολιτικών ελευθεριών δηλαδή να εμπλακούμε και να συμμετάσχουμε στην υπόθεση αυτή. Επίσης δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται με τον όρο εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να αρθεί το καθεστώς της απελευθέρωσης από τη θεώρηση. Τι εννοείται ακριβώς, τι σημαίνει αυτό. Μαζικές ροές, τι πώς ορίζεται το μαζικός ή τι άλλο μπορεί να σημαίνουν ροές. Και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με ε, τους εταίρους με τους οποίους έχουμε την υποχρέωση βίζας, θα ανοίξει πάλι το θέμα, θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις και το καθεξής. Βλέπω επίση ότι θέλετε να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να επανεισαγάγουν του ελέγχου στα ιστορικά σύνορα σε περίπτωση άκρο εξαιρετικών περιστάσεων κ.ο.κ. Αλλά από την άλλη μεριά θέλετε αυτό να το εντάξετε σε μια ε, κοινοτική διάσταση. Ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν από μόνο του, αλλά ταυτόχρονα θα αποφασίσει και η κοινοτική διάσταση. Τι σημαίνει αυτό. και πώς ορίζονται οι έκτακτες ε, περιπτώσεις ή η ίστατη ανάγκη. Επίσης βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό καθυστερήσεις. Ε, δεν θα θέλαμε λοιπόν ε, κάποιοι μετανάστες να περνούν από ελέγχους τόσο αραλυτικούς και διεξοδικούς που τελικά να γίνονται διάφανοι σαν, τη, την μέδουσα όταν περνούν από τα σύνορα, δηλαδή να πρέπει να, να εκθέτουν όλους την προσωπική ζωή. Ο κύριος Κοέλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε, που παρουσιάσατε τις καινούργιες σας πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε που επιτρέπετε στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στη διαμόρφωση αυτών των πρωτοβουλειών πριν τις παρουσιάσετε δημοσίως. Αλλά κυρίως σας ευχαριστώ για την ισχυρή σας αντίθεση και αντίσταση στην πρωτοβουλία ορισμένων κρατών μελών να αλλάξουν την νομική βάση και να αποφύγουν την συναπόφαση με το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση του, της λειτουργίας της Σέγγεν. Η Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντική, το είπατε και εδώ και στο Στρασβούργο. Χρειάζεται ένας καινούργιος μηχανισμός για την αξιολόγηση της Σέγγεν και χρειάζεται επίσης και ένα κοινοτικό σύστημα και για τους μάλλον ακόμα και για τις ε, αποφάσεις ε, προσωρινής ε, επιστροφής στους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα ευθυγραμμιζόμαστε. Ένα μόνο ερώτημα έχω σχετικά με τη Σέγγεν για το SIS 2. Όπως γνωρίζω, ε, προσωπικό μετακινήθηκε από το SIS2 στο VIS, στο Visa Information System. Ε, κάτι όμως που δημιουργεί κίνδυνο για περισσότερες ε, καθυστερήσεις στο SIS2. Ο κύριος Τζακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ντεμέρα επανειλημμένα την ευχαρίστηση για όλα αυτά που έκανε, ό,τι ήταν δυνατόν, για ό,τι ήταν δυνατόν την ευχαριστεί, δεν θα επαναλάβω στις ευχαριστίες. Συμφωνώ απόλυτα με αυτές τις εκτιμήσεις αξιολογήσεις. Η δεύτερη ανακοίνωση που, που μας παρουσιάσατε σήμερα έχει προφανή λόγο ύπαρξης, έτσι. Να δώσει συνέχεια στην πρώτη, θέτοντας στο επίκεντρο την αλληλεγγύη πριν μπείτε μέσω μιας μελέτης επιστημονικής πάρα πολύ σημαντικής αντιμετωπίσαμε το θέμα πριν από 20 χρόνια και περισσότερο έπεσε το τείχος. Εδώ και μερικέ μήνε έπεσε άλλο, άλλο τείχος, φράγμα στην ε, Μεσόγειο. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία έναντι των συνοριακών χωρών, έναντι αν θέλετε των παραμεθωριών χωρών, των χωρών που είναι στα νότια της Μεσογείου. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, Μέθοδο ε, ε, συλλογική. Ανεπαρκή είναι η πόρη όμω και χρειάζεται να προωθηθεί η κινητικότητα διότι η Ευρώπη μπορεί να χρειάζεται ανθρώπινους πόρους που προέρχονται από την Βόρεια Αφρική, από τον νότο της ε, Μεσογείου. Ε, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο ελπίζω. Αν η λιλεγγύη είναι κρίσιμης σημασίας, όπως σωστά εσείς είπατε και σήμερα, πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτή εν ώψη των νέων δημοσιονομικών προπτικών ούτως ώστε να δοθεί συγκεκριμένη υποστήριξη μέσω μεγαλύτερων οικονομικών, τεχνικών πόρων όφελος στι χώρε που εκτίθεται περισσότερο στις μεταναστευτικές ροέ, Διαφορετικά η λιλεγγύη την οποία συζητήσαμε και για την οποία εργάζεστε εσεί και σας το αναγνωρίζω, ίσως ε, να μην ανταποκριθεί στο στόχο που έχουμε θέσει αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 77 και 80 της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ρομέρο έχει το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Μάλστρομ. Ίσως δεν έχει υπογραμμιστεί αρκετά στη συζήτησή μας το εξής. Όταν μιλάμε για μεταναστεύσεις και αναμειγνύουμε την νόμη μετανάστευση και την παράτη μετανάστευση, λαθρομετανάστευση με θέματα ασύλου, ε, μπερδευόμαστε, διότι τα δύο αυτά προβλήματα μετανάστευση και ασύλου είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Στην ανακοίνωση για την μετανάστευση, το, η λέξη άσυλο εμφανίζεται μόνο στους πίνακε, πουθενά αλλού. Ακόμα και όταν μιλούμε για τι οδηγίε του πακέτου ασύλου, είναι ένα σύμπτωμα. Αυτό που συνέβη στη Βόρεια Αφρική είναι ε, κάτι έκτακτο, παρόλο ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Και η Ευρώπη απέδειξε ότι δεν διαθέτει μηχανισμό για την εντόπιση τέτοιων καταστάσεων. Ίσως εξαιτία της κακής διαχείρισης του θέματος από δύο κυβερνήσεις. Η εικόνα της Σέγγεν, η οποία προκύπτει όμως, ε, είναι πάρα πολύ αρνητική για όλους, διότι δείχνει σαν να μην υπάρχει καθόλου συνεργασία κοιτώντα την κατάσταση από την άλλη πλευρά, από την άλλη όχθη τη Μεσογείου, ενίσχυση του Σέγγεν σημαίνει ενίσχυση των συνόρων. Η Αίγυπτος και η Τινησία όμως δέχονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες, πολλές χιλιάδες ετούντων άσυλο που ε, προέρχονται από τη συγκρούση στη Λιβύη. Η Ευρώπη ενώ, ενώπιον αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να αντιδρά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε θέμα εικόνας μας, εξωτερικής μας εικόνας προς αυτές τις χώρες. Χρειάζονται να βρούμε καλύτερους τρόπους ε, να διαχειριστούμε την λαθρομετανάστευση και να μην μπερδεύουμε το θέμα της λαθρομετανάστευσης με το θέμα των ετούντων τον άσυλο. Στην Ελλάδα είδαμε πώς προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα και χρειάζεται πολύ περισσότερη χρηματοδότηση για να διαθέτουμε μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης που θα μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στους ετούντες άσυλο και τους λαθρομετανάστες. Χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια. Και στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων έχουμε φτάσει σε παράνοια. Διότι έρχεται ένας καθηγητής που έρχεται να να κάνει μια ομιλία σε ένα ε, πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Ή εμπειρογνώμονες, δικηγόροι, ε, επιστήμονες, ε, άνθρωποι ηλικιωμένοι 70 ετών που τους δεν του δίνουν θεώρηση γιατί λέει φοβούνται ότι θα δουλέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μείνουν εδώ να δουλέψουν. Είναι παρανοϊκή η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να διαπραγματευτούμε συμφωνίες επανεισδοχής όταν η εικόνα είναι τόσο μαυρωμένη. Ευχαριστώ. Η κυρία Εντβέλτ έχει το λόγο, όχι. Όχι, οπότε, εν τη αυτή περίπτωση, στην κυρία Σαρτζεντίνη πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Το περασμένο καλοκαίρι συζητήσαμε την κατάσταση με τις πρόσφυγες από την Ερυθρέα στην ε, Λιβική έρημο, που απειλεί το ότι θα αποσταλούν πίσω στην Ερυθρέα. Τώρα θέλω να μιλήσω για κατοίκους Ερυθρέας της Σομαλίας, και άλλους υπηκόους χωρών της ε, Αφρικής στην έρημο του Σινά, που είναι μεταξύ Αιγύπτου και Παλαιστίνης και Ισραήλ. Επεξεργάζεται το πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας σε συζητήσεις με την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο πρόσφυγες στην Αίγυπτο που ξεφεύγουν από τη Λιβύη και πάνε στην Αίγυπτο και ίσως θέλουν να τα καταφέρουν και να περάσουν τη Μεσόγειο και να πάνε στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή για δικό τους λόγο και πάνε προς το Ισραήλ. Από την Υποσαχάρη Αφρική πάνε στο Ισραήλ. Και υπάρχουν έμποροι ανθρώπων εκεί που δεν βγάζουν απλώς κέρδος από αυτούς τους ανθρώπους, όπως κάνουν συνήθως αυτοί, αλλά τους σκοτώνουν τους κρατούν ομήρους για πολύ περισσότερο. Τους δίνουν δορυφορικό τηλέφωνο μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή με την οικογένειά τους για να πάρουν περισσότερα χρήματα και αν δεν πληρώσουν δεν φτάνουν ποτέ στο Ισραήλ. Τους σκοτώνουν. Ο αριθμός των γυναικών που ζητούν άμβλωση από τη στιγμή που φτάνουν στο Ισραήλ είναι τεράστιος. Και αυτό διότι ευδιάστησαν καθοδόν και έμειναν επί στην έρημο του Σινά. Και το αγνοεί αυτό η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον η περασμένη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αν υπογράψουμε ένα πρόγραμμα περιφερειακής προστασία με την Αίγυπτο που θα καλύπτει τα θέματα μετανάστευση και ασύλου, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να πάνε εκεί και να εφαρμόσουν το κράτος δικαίου στο ΣΥΝΑ, διότι διαφορετικά η εκμετάλλευση των προσφύγων από την υποσαχάρια ε, Αφρική που πηγαίνουν στο Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Και δεν μπορούμε να υπογράψουμε πρόγραμμα προστασίας ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο με την Αίγυπτο για μετανάστευση και άσυλο χωρίς να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ λέω ο Πρόεδρος. κυρία Ένστ. Δύο πράγματα. Καταρχά, το ζήτημα των ελέγχων στα σύνορα. Θα ήθελα πολύ συγκεκριμένε απαντήσει και κάνω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Διαφάζω λοιπόν καταρχά ότι υπό ορισμένε συνθήκε μπορεί να προβλεφθεί μια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει κατόπιν λήψη σε αποφάσεω σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί ποια θα είναι τα κράτη-μέλη για τα οποία θα ισχύσουν εξαιρέσει. Δηλαδή θα επανεισαχθούν οι έλεγχοι. Ε, η ερώτησή μου είναι εξή. Είναι η απόφαση αυτή, η μελέτη αυτή έχει γίνει κατά τρόπο διαρθρωμένο, δηλαδή σκέφτεσαι ότι όντω μπορεί να υπάρξουν κράτη-μέλη τα οποία μπορούν μεμονωμένα να επανεισαγάγουν του ελέγχου ή θέλετε να διευκολύνετε την εισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα. Θέλετε να διευκολύνετε ή να καταστήσετε πιο δύσκολη την εισαγωγή των ελέγχων. Τι σημαίνει εξαιρετικέ περιστάσει. Για μένα, εξαίρεση μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή. Εξαίρεση μπορεί να είναι όμω επίση μεταναστευτικέ ροέ μαζικές μεταναστευτικέ ροέ. Μπορεί να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή ω φαινόμενο, αλλά ενδέχεται κάποια στιγμή να εμφανιστούν. Άλλο, άλλη περίπτωση. Ένα τμήμα των συνόρων να σημειώνει μεγάλη ε, προσέλευση, ε, μάλλον πολλά, πολλά αριθμα φαινόμενα ε, κλοπών. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Πώς το ορίζουμε και πώς τοποθετούμαστε μέσα σε όλο αυτόν τον προβληματισμό. Δεν βλέπω τι στόχο ακριβώς επιδιώκεται και ως εκ τούτου δεν βλέπω ακριβώς τι σημαίνει εξαιρετική περίσταση. Αυτή η ρήτρα της εξαίρεσης, ότι μπορεί δηλαδή ως ίστατη λύση και τα λοιπά, διασφαλιστική δικλίδα ή για λόγους ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό, σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύει και επίσης για το Smart Border. Είπατε ότι εισάγεται ή πρόκειται να εισαχθεί μια νέα τεχνολογία για την οποία θα ήθελα να μα πείτε δύο λόγια παραπάνω. Τι εννοείται ακριβώς νέα τεχνολογία. Ευχαριστώ. Κύριε Παρικολάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτροπέ, που είστε εδώ μαζί μας μία ακόμα φορά. Στο πρόσφατο παρελθόν ε, υπογράφηκαν διμερείς ε, συμφωνίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα με τρίτες χώρες όπως το Μαρόκο, τη Λιβύη, την Τινησία κλπ. Με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και με κάποιο τρόπο καταφέραμε να ελέγξουμε τις ροές των λαθρομεταναστών τα τελευταία χρόνια. Τώρα βέβαια η κατάσταση άλλαξε. Οπότε η ερώτηση είναι η εξή. αυτές οι ε, εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας, τις οποίες αναφέρατε, αποτελούν προετοιμασία για ένα καινούριο πλαίσιο επανεισδοχής ε, με αυτές τις χώρες και κάτι που συνδέεται με αυτό. εξακολουθούμε να παρατηρούμε τεράστια είσοδο ε, μεταναστών από την Τουρκία. Ε, καταφέρατε να υπογράψετε τη, μια συμφωνία με την Τουρκία, το Συμβούλιο τη δέχτηκε, αλλά η πραγματικότητα είναι η εξή. Προκειμένου να δεχτεί η Τουρκία την επανεισδοχή ε, τρίτων χωρών στην επικράτειά της, ε, ε, επέβαλε μια, ένα όρο αυτό να ξεκινήσει τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύω της συμφωνίας. Δύο χρόνια λοιπόν μέχρι την έναρξη ισχύω και άλλα τρία χρόνια πέντε μέχρι ότου η Τουρκία να δεχτεί το 90% των ε, λαθρομεταναστών φτάνουν στο 2016-2017. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί με την Τουρκία και να συνδυάσετε τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία, γιατί δίνουμε στην Τουρκία εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τα σύνορα της και τους σύνορακούς ελέγχους. Να συνδυάσουμε λοιπόν αυτή τη χρηματοδότηση με την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής. Ευχαριστώ, κ. Δεγιόντ. Ένας από τους, μία από τους συναδέλφους είπε ότι ε, εκπλήσεται που βλέπει την κυρία Μάλστρομ να αντιμετωπίζει επίσης την διαφθορά. Εμένα με χαροποιεί αυτό. Και πολλοί ε, μαζί με μένα υπέγραψαν ένα σημείο που τη στείλαμε για αυτό το θέμα. Ε, σήμερα η διεθνής διαφάνεια ε, δημοσιοποίησε ε, τι, πέντε εκθέσεις για την εφαρμογή της σύμβασης του ε, ΟΑΣΕ ε, από διάφορα κράτη-μέλη. Τα μισά τουλάχιστον κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν επαρκώς τη σύμβαση αυτή. Συνεπώς αναμένουμε βέβαια το, την ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά επιπλέον δεν πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι είναι επίγον Δεδομένου πολλέ πολλές εταιρείε τιμωρούνται από κράτη-μέλη, ενώ κάποιε άλλε δεν τιμωρούνται καθόλου. Όπω για παράδειγμα την Philips, η Philips στην Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν παίρνει καθόλου πρωτοβουλίε για αυτό το ζήτημα, ενώ η Πολωνία ε, για την ίδια εταιρεία ε, επιβάλλει ποινέ. Συνεπώς δεν είναι επίγον να επιβληθεί, να εφαρμοστεί η ίδια νομοθεσία για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουμε μια διαδικασία fast track ενδεχομένως για την εφαρμογή της σύμβασης του ΑΣΕ. Και ενδεχομένως να υιοθετήσουμε, να θεσπίσουμε και ε, κάποιο είδους ε, μέσο ή μέτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η εφαρμογή να γίνει με ομοιόμορφο τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτό το μήνυμα στον έξω κόσμο. Περιμένω βέβαια το, την ανακοίνωση επιτροπή, αλλά έχω την εντύπωση ότι το θέμα είναι πιο επίγον από ό,τι νομίζαμε. Van de ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Η ερώτησή μου ε, σχετίζεται με την ερώτηση της κυρίας Βαζόν και της κυρίας Κέλλερ. Ίσως έχουμε διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, αλλά το θέμα είναι το ίδιο. Μπορούν ορισμένα κράτη-μέλη δηλαδή να εισαγάγουν την υποχρέωση για θεώρηση. Φερρυπίν έναντι τη Αλβανία ή τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ή εν τέλει είναι απαραίτητη η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον τύπο στις κάτω χώρες. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η κατάσταση. Και επίσης θα ήθελα προκαταβολικά να στήσω συγγνώμη, δεν θα μπορέσω να ε, μείνω να ακούσω την απάντησή σας, αλλά ή, ε, το προσωπικό μου, οι συνεργάτες μου θα μείνουν για να σημειώσουν τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την ε, αθρώα συμμετοχή τις πολυάριθμε ερωτήσει, αλλά και το χρόνο που αφήσατε ελεύθερο για να δώσει απαντήσει η Επίτροπο Μάλστρομ, που ξαναπαίρνει το λόγο. Είχατε αισθήσει το λόγο, κύριε Μίλντερ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά... Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ε, θα έχουμε και τους συντονιστές μετά ο πέρα τη παρεμβάσεω τη Επιτρόπου και θα την ευχαριστώ προκαταβολικά εάν εξοικονομήσει λίγο χρόνο ώστε να ξαναπάρουμε την συνεδρία στα χέρια μα με του συντονιστέ. Ναι, Πρόεδρε. Ε, Σα διαβεβαιώ, λέει ο κύριο Μίλτερ, ότι είχα στήσει το λόγο και είδα και κάποιον να μου λέει ναι, ναι, σε σημείο. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Ε, πρέπει να σημειώσω ότι έχει δώσει σημασία στην Επιτροπή μας και έχει προσελκύσει σημασία, έχει προσελκύσει ενδιαφέρον η παρουσίαση εδώ, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλου επιτρόπου τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι η κυβέρνηση Ολλανδίας έχει εισαγάγει κάποιες ομάδες ελέγχου αντίστοιχες με αυτές που έχει η Δανία και ότι προσπαθεί να επανεισαγάγει του ελέγχου. Έχει υπόψη τη Επιτροπή κάτι τέτοιο. Ε, δεύτερον, σε σχέση με την ε, Δανία, είναι πολύ αρνητική η στάση της Επιτροπής, αλλά τι χρονοδιάγραμμα σκοπεύει να ακολουθήσει η Επιτροπή, ε, περιμένει τις απαντήσεις της Δανίας και μετά τι μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε. Ευχαριστώ η Επίτροπος παρακαλώ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ξεκινήσω με την κυρία Φαζούν. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εισαγάγουν μόνα του. Έχουμε μια κοινή πολιτική για τη βίζα και ω εκ τούτου δεν μπορεί κανεί να λάβει μονομένε αποφάσει. Δεν υπάρχει αυτοματοποίηση δηλαδή η αυτόματη εισαγωγή. Πολλέ είναι οι διαδικασίε που θα χρειαστεί να ακολουθήσει κάποιο κράτο μέλο. Θα τα δούμε ε, όπως άλλωστε τώρα βλέπουμε και με τη Μακεδονία και τη Σερβία το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να εμποδίσουμε ενδεχόμενες καταστρατηγήσεις του δικαίου. Δυστυχώ, όμω βλέπουμε ότι υπάρχουν καθημερινά κάποια προβλήματα τέτοιου τύπου από ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης, το σύστημα ε, έγκαιρης προειδοποίησης θα φροντίσουμε να εισαγάγουμε, έτσι ώστε να έχουμε πράγματι ως πράγματι τελική ε, έσχατη λύση την υπαρισαγωγή των ε, ελέγχων ή τη βάλω την υπαρισαγωγή των θεωρήσεων. Το Κοινοβούλιο φυσικά μπορεί πάντοτε να προσκαλεί την Επιτροπή για συζήτηση θεμάτων που το ενδιαφέρουν ως προς τις εκτελεστικές εξουσίες για την ε, κύριε Λάντφορντ. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση σχετική με τη λέξη. Ε, σε μια συνέντευξη τύπου, αν δεν απατώμε, τοποθετήθηκα και έχει καταγραφεί. Σαφώς είπα ότι μπορεί ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιπλέον των μηχανισμού ε, αξιολόγησης, διαδικασία με τα κράτη-μέλη, λοιπά, μέσα οι διευκρινήσεις, ε, κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή όλα αυτά καθιστούν πολύ πιο, γρήγορο, πιο δύσκολο για τα κράτη-μέλη μονομερώς να εισαγάγουν. Αυτό θέλουμε. Να αποφύγουμε το ε, φαινόμενο κάποιο κράτος μέλος μεμονωμένα να κάνει. Βέβαια ε, μπορεί με μια εξαιρετική περίσταση, φερειπίν μια τρομοκρατική ε, επίθεση, μεμονωμένη, σημαντική να χρειαστεί. Πάντως εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό στο δυνατόν πιο δύσκολο, ε, τουλάχιστον ε, όσον αφορά τη μόνιμη μορφή του. Δηλαδή, μπορεί μεν περιστασιακή έλεγχη σύντομη διάρκεια, φερρυπίν έλεγχη ε, για να αποτρέψουμε το φαινόμενο του χουλιγκανισμού σε πούλμαν ή σε, σε λεωφορεία που έρχονται από τη μια χώρα στην άλλη. Τότε ναι, καταλαβαίνω, για μια, δύο μέρε, τρει μέρε. Αλλά σε μια πιο μόνιμη μορφή πρέπει η διαδικασία να είναι πιο περιπλοκή και πιο εμπεριστατωμένη. Η, διαδικασία στη, κατάσταση στη Βόρεια Αφρική υπόθηκε από την κυρία Κέλλερ και από άλλου ότι ναι, πιέζει πολύ το σύστημά μα, επιβάλλει πολλέ πιέσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να αποστείλουμε το μήνυμα πόσο εκ τούτου αλλάζουμε το Σέγγεν. Κυρία Ρομέρο, νομίζω ότι απευθύνετε τους, ε, την οργή σα, ε, αποστέλλετε την οργή σα προ το εσφαλμένο θεσμικό όργανο. Το ότι υπάρχουν προβλήματα στην Νότια Μεσόγειο δεν σημαίνει ότι ε, πρέπει να καταργηθεί το Σέγγεν ή να αποδυναμωθεί. Από τις ε, πολλέ εκατοντάδε χιλιάδων που έχουν αποχωρήσει από τη Λιβύη, λίγοι είναι αυτοί, ελάχιστοι είναι αυτοί που ήρθαν στα ε, κράτη της Ευρώπης. Φυσικά δεν υποτιμώ τη σημασία των μεταναστευτικών ροών προς την Ιταλία και τη Μάλτα, αλλά συνολικά, γιατί βέβαια εκεί έπεσαν πολλά ε, πολλοί μετανάστες ταυτόχρονα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά συνολικά και σε βάθος χρόνου ε, μετανάστες από την νότια όχθη της Ευρώπης δεν ήταν τόσο πολλοί. 323 ήταν εκείνοι της Μάλτας και 800 του UNHCR. Από τα 27 κράτη-μέλη, 800 συνολικά μετανάστες ή πρόσφυγες δεν είναι πολλοί. Είναι μάλλον λίγοι. Η κυρία Κέλλερ, ναι, για την θεώρηση στο διαβατήριο φυσικά δεν πρόκειται για επαναδιαπραγμάτευση. Έχουμε έναν μηχανισμό που έχει θεσπιστεί και ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν. Κύριε Κουέλο, οποιαδήποτε ε, ανάθεση ή τοποθέτηση προσωπικού γίνεται από τις σχετικές υπηρεσίες. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να πω για τις τεχνολογικές εξελίξεις τα πράγματα πάνε πολύ καλά, πλην όμως υπάρχει η πρόκληση να είναι εγκαίρως έτοιμα τα κράτη-μέλη με την επάνδρωση που χρειάζονται, με τον ε, ανθρώπινο δηλαδή, με το ανθρώπινο δυναμικό που θα υπάρχει. Επίσης δεν έχω ακούσει να υπάρχει πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθώ το θέμα τακτικά και αν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ασφαλώς θα το είχα ακούσει. Κύριε Ιακολίνο, χρηματοδότηση. Οι συνάδελφοί μου θα σας ε, παρουσιάσουν αύριο το έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, όπου καλύπτεται και το θέμα των κονδυλίων, των μέσων που διατίθενται στην γειτονία μας προς τον Νότο, αλλά και την Ανατολική γειτονία. Τα σχετικά κονδύλια λοιπόν, και πρέπει να πω ότι υπό τη δική μου ευθύνη, και σας το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω, θα προσπαθήσω να διευκολύνω τη χρήση αυτών των κονδυλίων, ώστε να μπορούμε να τα ε, συνδυάσουμε. Για αυτή τη στιγμή υπάρχει έω και επικάλυψη. Πάντω μπορείτε να στηρίζετε σε μένα, όπω και εγώ στηρίζομαι στη βοήθεια του Κοινοβουλίου, που στο δικό μου τομέα αρμοδιοτήτων θα υπάρξει αυτή η ε, αποτελεσματική χρήση και πάντω όχι μείωση των κονδυλίων. Αντίθετο, θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν προσθέτει προστιθέμενη αξία στον χώρο τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών. Κύριε Αργεντίνη ε, εν γνώση των προβλημάτων που επισημαίνεται ε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η κυρία Άστον βεβαίω είναι ενήμερη για το θέμα και όλο ο ε, διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από την κινητικότητα, από την ασφάλεια, τη μετανάστευση έχει να κάνει ακριβώ με την ιδέα του ασύλου, την προσφορά ενό συστήματο ασύλου ε, συμβατού βέβαια με τα διεθνή ε, με τι διεθνεί προδιαγραφέ. Και αυτό το συζήτησα στο Κάιρο την, στην τελευταία μου επίσκεψη με τον Υπουργό των Εσωτερικών. Είμαστε ενήμεροι για τα προβλήματα που επισημαίνετε, κυρία Σαρτσεντίνη, και θα τα παρακολουθούμε διαρκώ. Ε, νέα τεχνολογία, smart borders. Ναι, μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα, αλλά κάποιο ο οποίο διασχίζει τα σύνορα καθημερινά ενδεχομένω για λόγου επαγγελματικού ε, ή σπουδαστέ φερρυπίν, όπου ε, έχουν δεδομένη ε, την νόμιμη αυτή δυνατότητα, μπορεί να υπάρχει ένα είδος token, ένα είδος δηλαδή μικρομηχανήματος, το οποίο θα τους επιτρέπει να περνάνε γρήγορα με μια μαγνητική κάρτα ενδεχομένως ε, χωρίς ταλαιπωρία τα σύνορα. Επίσης ευχαριστώ πολύ για τις συστάσεις και παρατηρήσεις για, τη διεθνή, για, το Amnesty, για το Amnesty International Διεθνή Αμνηστία και τις λοιπές προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ, θα τις λάβουμε υπόψη για την επανεισδοχή. Ε, όντως, εν γέννη, και αυτό νομίζω το είχαμε επισημάνει και στην παρουσίαση που σας ε, είχαμε κάνει πρόσφατα, η επανεισδοχή θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε από τρίτε χώρε να επανεισδέχονται ή να δέχονται και πάλι σκόλπου του κάποιου, ε, εάν δεν έχει γίνει ευρύτερη συζήτηση για το ε, για τη διαχείριση των συνόρων. Το θέμα, ας πούμε, της ε, απαλλαγής από τη θέωση των διαβατηρίων ισχύει για άλλες χώρες, δεν ισχύει για την ε, Τουρκία. Δεν το έχουμε συζητήσει μαζί τους και ως εκ τούτου και εκείνοι δεν υπογράφουν τη Συμφωνία Επανιστοχής γιατί θεωρούν ότι θα έχουν δικαίωμα στην απαλλαγή από τη θεώρηση διαβατηρίου. Είναι και υποψήφια χώρα και συμφωνώ, έχουν δίκιο σε αυτό που λένε τώρα. Όπως ξέρετε, η Τουρκία έχει μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία και ελπίζουμε ότι μετά από αυτήν θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει στο πρόβλημα. Για τον κύριο Μιούλτερ. Χρονοδιάγραμμα. Είχαμε ζητήσει διευκρινήσει από την ε, Γαλλία, την Ιταλία, τη Δανία και πιστεύω ότι και με, τους, ε, με τις κάτω χώρες που θα συζητήσουμε αύριο θα έχουμε ε, συζητήσει και διευκρίνηση των θεμάτων αυτών. Την Παρασκευή, αν δεν απατώμενη σειρά τη Δανία. Τα παρακολουθούμε λοιπόν τα θέματα. Ε, χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχουμε πει ότι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία θα λάβουμε κάποιε συγκεκριμένε αποφάσει. Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά ήταν όλα. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την Επίτροπο Μάλστρομ για τι προσπάθειε τη. Μα βοηθάτε πολύ. Βοηθάτε πολύ την Επιτροπή μα στην επιτέλεση του έργου της όχι μόνο λόγω της συχνότητας αλλά και της έντασης και της καλής διάθεσης για συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε για πέντε λεπτά και ξαναρχίσουμε με τους συντονιστές και κλεισμένο των θυρών.